Ladies and gentlemen, please be seated. We start immediately. Λοιπόν, αρχίσουμε αμέσως. Τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Λοιπόν, πρώτο θέμα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να σας ενημερώσω ότι η προτεραιότητα για τη διερμηνία είναι οι γλώσσες των, των τακτικών μελών της Επιτροπής μας, συμπληρωματικά για το σημείο της ημερήσιας διάταξης για την Κρυμαία. Έχουμε διερμηνία στα ρωσικά. Οπότε θα έχετε δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη διερμηνία από αυτή τη γλώσσα. Η διερμηνία μας επίσης μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Και αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, να περάσουμε στο επόμενο θέμα της μέρης της Και θεωρώ ότι εγκρίθηκε η Μέρες διάταξη. Κυρίες και κύριοι, Σήμερα κλείνει περίπου χρόνος από την απαράδεκτη και παράνομη προσάρτηση, όπως γράφουμε σε όλα μας τα έγγραφα, της Κρυμαίας από την Ρωσική Ομοσπονδία. Και γι' αυτό θα ασχοληθούμε ως πρώτο θέμα της ε, ημερήσιας διαταξής μας με αυτό το θέμα. Και έχω τη χαρά να καλωσορίσω κάτι συνεδρίαση την αυτοεξοχότητα των πρέσβη της Ουκρανίας, τον οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά, όχι μόνο στην Επιτροπή μας ΣΕΝΤΕ, αλλά και στην Επιτροπή ΑΦΕΤ εξωτερικών σχέσεων, είναι ο κύριος Κανσταντίν Ελισέριεφ. Επίσης έχουμε τον ηγέτη του Κοινοβουλίου των Τατάρων της Κρυμαίας, του Μετζλής, είναι ο κύριος Ρεφάτ Τσουμπάροφ. Τον έχουμε ήδη συναντήσει στις Βρυξέλλες, ορισμένα μέλη της Επιτροπής μας, κατά την ε, πρόσφατη αποστολή μας στο Κίεβο. Επίσης τον συναντήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις. Αυτό το θέμα το συζητάμε σε συνδυασμό με την ε, κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας και καλωσορίζω τον κύριο Αντζέι Πλένκοβιτς που είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας αυτής που όπως ε, σχεδόν σε όλες τις ε, συνεδριάσεις μας όπου συναντηθήκαμε με εκπροσώπους ε, της Ουκρανίας είναι και σήμερα μαζί μας και θα ανταλλάξουμε απόψεις για την επίσκεψη στην ε, Ουκρανία αργότερα. Επίσης έχουμε προσκαλέσει έχουμε προσκαλέσει μέλη της Υποεπιτροπής ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ορίζω τον εξοχόγατο αρχιεπίσκοπο της ε, Κρυμαίας, τον Ουκρανό Ορθόδοξο αρχιεπίσκοπο της ε, Κρυμαίας, Κλίμεντα, και επίσης τον αρχιεπίσκοπο του Τσέρνιχιφ, της Ουκρανικής ε, Ορθόδοξης Εκκλησίας, που εκπροσωπεί το Πανουκρανικό Συμβούλιο Εκκλησιών, που εκπροσωπείται στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς από εκείνον. Είναι εδώ παρόντες για να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με τους ευρωβουλευτές. Καλωσορίζω επίσης τον εξέχοντα δήμονα που έχει παίξει την εξέχουσα κυρία Ιρίνα Μπρουνόβα Καλισέτσκαγιά, που έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Επειδή ο κύριος Πλένκοβιτς όμως πρέπει να φύγει, να του δώσω ε, πρώτα το λόγο σε εκείνον. Ευχαριστώ κυρία Φωτζίγκα, κύριε Πρέσβη, κύριε Τσουμπάροφ, κύριε Πρόεδρε του Ματσλής, ε, κύριε Αρχιεπίσκοπη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εμπειρογνώμονες. Είναι μεγάλη χαρά που μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ της ΣΕΝΤΕ και της αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Ουκρανία. Για την Κρυμαία. Κλείνει χρόνος από την παράνομη και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο προσάρτηση αυτού του σαφούς ουκρανικού εδάφους από τη Ρωσία. Ήδη το Δεκέμβριο αποκινούμε την αντιπροσωπεία και την υποεπιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα συζητήσαμε την κατάσταση στην Κρυμαία, τις διάφορες ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα δεινά που υφίστανται οι κάτοικοι της Κρεμαίας, άρα και οι τάταρ της Κρεμαίας, μαζί με τον κύριο Τσουμπάροφ. Και επίσης ε, στη συζήτηση που κάναμε πριν από ένα χρόνο καταδικάσαμε σαφώς την προσάρτηση αυτή και επαναλάβαμε την πολιτική μη αναγνώριση αυτού του τετελεσμένου γεγονότος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην Ουκρανία, στο Κίεβο, πολύ πρόσφατα συζητήσαμε την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στην Κρυμαία με τους συνομιλητές μας και θεωρούμε ότι όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος δεν έχει ξεχάσει και δεν θα ξεχάσει την κατάσταση στην Κρυμαία και τα δεινά του λαού της. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συζήτησή μας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους Ουκρανούς φίλους μας, το λαό της Κρυμαίας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα παράνομα, παρανόμως κατεχόμενα δάφη του Ντανμπάς θα επανέλθουν στην ε, Ουκρανία αλλά και η Κρυμαία θα επανέλθει στην Ουκρανία όπου ανήκει. Ευχαριστώ κύριε Πλένκοβιτς και τώρα έχετε το λόγο ε, εξοχότατε. Ευχαριστώ κύριε Φωτίγκα αξιότιμα μέλη, κύριε Πλέγκοβιτ, ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτή του ειδικού, της ειδικής εκδήλωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς, όπως σωστά είπατε, αυτή η συζήτηση διεξάγεται ένα χρόνο ακριβώ μετά την παράνομη προσάρτηση της Ουκρανίας. Θέλω να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Τσούμπαροφ, τον Αρχιεπίσκοπα Κλίμεντα και την κυρία Ειρήνα που ήρθαν στι Βρυξέλλε παρά το πόσο πολύ άσχολοι είναι. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δυνατότητα που μας δίνεται για να ενημερωθούμε, να άλληλο ενημερωθούμε από πρώτο χέρι για την κατάσταση στην Κρυμαία. Η συνάντηση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις της προσάρτησης της Κρυμαίας. Τι διαπιστώνουμε στην Κρυμαία τώρα. Κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπίεση και την στρατιωτικοποίηση της Κρυμαίας. Αυτό είναι η ρωσική ειρήνη, Ρούσκι Μύρ. Σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με το σαφές όνομα η Κρυμαία ταξίδι προς την μητέρα πατρίδα, ο πρόεδρος Πούτιν παραδέχθηκε ότι η Ρωσία ενορχίστρωσε άμεσα τα γεγονότα στην Κρυμαία. Ένα χρόνο το αρνούνταν. Τώρα επιτέλους το παραδέχονται. Παραδέχονται ότι επιθέσεις κατά της κυριαρχίας και αδεαφικής ακαιρότητας της χώρας μου προγραμματίστηκε εδώ και πολύ καιρό και διεξάχθη με πολύ συντονισμένο τρόπο. Αυτή είναι η πρώτη προσάρτηση εδάφους κυριάρχου κράτους στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η προσάρτηση αποτελεί τη σοβαρότερη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, το σοβαρότερο διεθνές έγκλημα, το οποίο το διέπραξε ένα κράτος που υποτίθεται ότι είναι θεματοφύλακας ε, της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσφατα έστειλα μια επιστολή στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καλώντας επιγόντως την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει σε αυτήν την ομολογία του Πρόεδρου Πούτιν. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι θα επαναβεβαιώσει την πολιτική της θέση για την Κρυμαία, αλλά επίσης θα εκφραστεί και νομικά για το θέμα αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο θέμα συνόρων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η προσάρτηση της Κρυμαίας επιτρέπει την επανεξέταση των συνόρων στην Ευρώπη, την Ασία, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Προφανώς η πολιτική της Ένωσης προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο αν επανέλθει η κυριαρχία επί της Κρυμαίας. Άρα πρέπει να περάσουμε σε υψηλότερο επίπεδο κυρώσεων και να μην αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κρυμαίας όπως δεν την αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο μόνος ειρηνικός τρόπος να επανέλθουμε στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας θα μας επιτρέψει να αποτρέψουμε ένα επικίνδυνο προηγούμενο στην παγκόσμια πολιτική δεν έχουμε δικαίωμα να επιτρέψουμε να θριαμβεύσει ο επεκτατισμός και η εκδικητικότητα. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δικαίωμα να επιτρέψουμε να θριαμβεύσει ο εμπεριαλισμός και ο επεκτατισμός. Αγαπητοί φίλοι, δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο. για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρεφά Τσουμπάρου θα πάρει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые члены Αξιότιμα μέλη της Υποεπιτροπής ε, για την ε, άμυνα Θα ήθελα πρώτα απ' όλα ως εκπρόσωπος των Μέτλη και των Τατάρων της Κρυμαίας να σας ευχαριστήσω για την προσοχή ε, που δείχνεται για την Κρυμαία μετά την ε, παράνομη προσάρτηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία πριν από ένα χρόνο της Χερσονήσου. Όπως είπε η Πρόεδρος, τις περασμένες εβδομάδες είχαμε άφθονες ευκαιρίες επαφών με τα μέλη της υποεπιτροπής σας για μια σειρά ζητημάτων. σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην Κρυμαία, την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πιθανές εξελίξεις. Αυτή ε, η σημερινή μας συνεδρία είναι η φυσική συνέχεια αυτού του διαλόγου. Τα όσα διαμήθησαν το 2014 τον Απρίλη και τον Μάη στον Τονέτσκ και στο Λουγκάνσκ οδήγησαν στον τραγικό θάνατο επίσης των 300 επιβατών του Boeing, του αεροσκάφους των Malaysian Airlines και οδήγησαν στη συνέχεια στην προσάρτηση της Κρυμαίας. Οι συμφωνίες Μίνσκ 1 και 2 δεν αναφέρονται την κατάσταση στην Κρυμαία και σε πολλές φορές όταν συζητούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τις μελλοντικές κυρώσεις όταν συζητούν για την επιβολή επιπρόσθετων κυρώσεων ή άρση των κυρώσεων ε, ε, συζητούν μόνο για, την, ε, για μία αίρεση, δηλαδή την σταθεροποίηση της ε, κατάστασης στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά δεν αναφέρονται καθόλου στην Κρυμαία. Με την ε, επέτειο, πολλά, πολλοί θεσμοί, ευρωπαϊκοί, το ΝΑΤΟ, αλλά και η διεθνή κοινότητα θα έπρεπε να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την Κρυμαία. Εάν δεν επιστρέψει στην επικράτεια της ε, Ουκρανίας ε, η Κρυμαία, δεν θα μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την ρωσική επιθετικότητα. Είμαστε πεπισμένοι πως είναι επιτακτική ανάγκη να αναλυθούν τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Λοιπόν, για την κατάσταση στην Κρυμαία έχει παρέλθει ήδη ένας χρόνος και δυστυχώς οι πλέον ζωφερές προβλέψεις μας έχουν επιβεβαιωθεί. Στην πρώτη φάση της κατοχής υπήρξαν υπερβολικές υποσχέσεις για την διαφύλαξη δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών από τις κατοχικές δυνάμεις. Μας υποσχέθηκαν οικονομική ευημερία και υψηλά πρότυπα για την οικονομία. Όμως, ε, ξανεμίστηκαν όλες αυτές οι υποσχέσεις ε, μέχρι το τέλος του 2014. Ένα μέρος του πληθυσμού πίστεψε τις ε, υποσχέσεις ε, των κατοχικών δυνάμεων στις υποσχέσεις της Μόσχας και ε, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κατασταλτικό μηχανισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας τον αδυσόπιτο αυτό μηχανισμό που διέψευσε τις υποσχέσεις Για ορισμένους βεβαίως υπήρξαν ναι, υψηλοί μισθοί και υψηλές συντάξεις για κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού. Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας, οι ερευνητικές επιτροπές, η εισαγγελία ήταν οι υπηρεσίες που έλαβαν τα περισσότερα κονδύλια διότι υποβάλλουν τακτικά αναφορές στη Ρωσία παρατηρήθηκαν φαινόμενα όπως ε, ε, εξαφανίσεις νέων τατάρων και ορισμένοι βρέθηκαν δολοφονημένοι στη συνέχεια πολλές συλλήψεις, ε, διώξεις ακτιβιστών από το κίνημα των Τατάρων, εκβιασμός, εκφοβισμός μελών των Μέιτσλης, των μελών των Μέιτσλης απαλωτρίωση ε, περιοσιακών στοιχείων των μέτλης και μη κυβερνητικών οργανώσεων ούτως ώστε να καταπατηθούν τα δικαιώματα και οι φιλοδοξίες των Τατάρων και άλλων εθνικών μειονοτήτων. Στην Κρυμαία υπάρχουν πολλές Δίκε σε σχέση με αυτά που έγιναν στις 26 Φεβρουαρίου του 2014 μεταξύ άλλων. Παρακαλώ να θυμηθείτε αυτήν την ημερομηνία 26 Δευτέρου 2014 παρά τις παρατηρήσεις του Προέδρου Πούτιν δεν μπορούμε να μιλήσουμε παρα, για παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι ε, Τατάροι τότε ε, ε, διοργάνωσαν ένα μαζικό συλλαλητήριο για να υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της Κρυμαίας και πολλοί τώρα διώκονται από πλευράς της Ομοσπονδιακής ε, Ομοσπονδίας Ασφαλείας FSB υπάρχουν βίντεο των γεγονότων του Φεβρουαρίου αλλά και του Ιανουαρίου και βάσει του ποινικού δικαίου της Ρωσίας πολλοί απειλούνται με δεκαετή κάθερξη. Ο Μούσταφα Τζαμιλέφ εκείνη την ημέρα προσπάθησε να μπει στην Ουκρανία από την ε, πυρωτική Ουκρανία και στο διοικητικό αυτό σύνορο ήρθαν να τον συναντήσουν πάνω από 2.500 ε, τατάροι της Κρυμαίας. Ε, δεν μπορέσαμε όμως να εξασφαλίσουμε ένα διάδρομο εισόδου για τον κύριο Τζεμίλοφ ε, λόγω της περιμέτρου των Ρώσων και όλοι όσοι συνελήφθησαν εκείνη την ημέρα διώκονται αυτή τη στιγμή και απειλούνται με αυτή τη δεκαετή κάθεξη που προανέφερα. Ήθελα δεν να τονίσω πως οι μελλοντικέ εξελίξεις θα είναι συνάρτηση μιας ε, σειράς ζητημάτων που σχετίζονται με τις ε, ρωσικές, ε, με τα όσα αποφασίζει και κάνει η Ρωσική Ομοσπονδία σε σχέση με την Κρυμαία. Ε, χρησιμοποιούνται μέσα από τους ευρωπαίους θεσμούς ε, για να αναχαιτιστεί, όπως έλεγα, η ρωσική επιθετικότητα και όσο συμβαίνει αυτό αναλαμβάνονται ολέδα και πιο κατασταλτικά μέτρα ε, επιτόπου. Οι τοπικές αρχές αναλαμβάνουν αυτά τα μέτρα εναντίον των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν ε, δίνεται άδεια διαμονής ε, για τους ε, Τατάρους. Έχουν κλείσει όλα τα σχολεία όπου διδάσκεται η γλώσσα μας. 14 σχολεία διδασκάν την γλώσσα μας στο παρελθόν και θα γίνει και μια εκδήλωση υπέρ του καναλιού ATR που μεταδίδει στην Ταταρική και από πρώτη Τετάρτου θα κλείσει, θα πάψει η λειτουργία του καναλιού μετά την απόφαση των αρχών. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και εν είδη συμπεράσματος ε, επιτρέψτε μου Να επαναλάβω τα όσα είπα και στην προηγούμενη σύσκεψή μας ότι ο πόλεμος ε, κατά της Ουκρανίας άρχισε με την προσάρτηση της Κρυμαίας και μόνο έτσι μπορεί να τελειώσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τσουμπάροφ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα μόνο ένα σχόλιο να κάνω για να εξηγήσω για ποιο λόγο προωθούμε και αναδεικνύουμε σε τόσο σημαντικό το ζήτημα των ε, Τατάρων της Κρυμαίας και κυρίως ως προς ε, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ο Βλαντιμίρ Πουτίν και το καθεστώς του Κρεμλίνου συνήθως μιλάουν για την πλειοψηφία των ρωσοφόνων στην Κρυμαία δικαιολογώντας ε, τη δράση τους. Ας θυμηθούμε όμως ότι ε, πριν από όχι τόσο πολύ καιρό έγινε πρώτα εθνική κάθαρση ε, με απέλαση των ε, Τατάρων Ε, οι οποίοι μετεκαταστάθηκαν σε διάφορα μέλη της πρώην ε, Σοβιετικής Ένωσης και στη συνέχεια άρχισαν να επιστρέφουν στα πάτρια μετά την ε, ανακήρυξη ανεξαρτησίας της Ουκρανίας και τώρα επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία για δεύτερη φορά. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε να συζητήσουμε και να προβάλλουμε ε, το θέμα των Τατάνους Κρυμαίας. τώρα θα ήθελα για τη συζήτηση να δώσω το λόγο στους βουλευτές. Ε, εάν έχουμε χρόνο στη συνέχεια θα ήθελα, αν συμφωνείτε, να ακούσουμε και τους αρχιεπισκόπους τους επίτιμους προσκεκλημένους μας. Αλλά αυτό μόνο κατόπιν συνένεσή σα και μόνο στο βαθμό που θα έχουμε βαθμό. Οι συντονιστές, ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη, κύριε Τσουμπάροφ για τις παρουσιάσεις σας. Την προηγούμενη εβδομάδα πήγαμε στο Κίεβο και όσοι πήγαμε σας έχουμε ήδη συναντήσει εκεί και συζητήσαμε την κατάσταση στην Κρυμαία και ιδιαίτερα την κατάσταση της εθνικής σας ομάδας η οποία είναι πολύ λυπηρή. Ηρωνικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι όμως και έκπληξη διότι όταν ο Πούτιν δεν χορηγεί ανθρώπινα δικαιώματα και παραποιεί την αλήθεια για ολόκληρο τον πληθυσμό του, γιατί να μην το κάνει και για αυτούς, είναι μια συστημικά αυταρχική κυβέρνηση. Επειδή σας έχουμε εδώ στην ε, υποεπιτροπή μας, ήθελα να θέσω το ερώτημα τι γνωρίζουμε για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που είναι παρούσες εκεί. Είναι αποδεκτή, είναι στο επίπεδο της συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τη Σεβαστούπολη ή όχι. Τι γνωρίζετε λοιπόν εσείς. Πόσες ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις υπάρχουν στην Κρυμαία, πού στρατοπεδεύουν είναι πιο πολύ προς το βορρά κοντά στην υπόλοιπη Ουκρανία. Έχουν καθόλου ατομικά όπλα ε, εγκαταστήσεις στην Κρυμαία. Γιατί υπάρχουν κάποιες τέτοιες αναφορές ή μάλιστα και απειλές από πλευράς Ρώσων. Πώς έχουν τα πράγματα. Και κάτι άλλο τα ρωσικά στρατεύματα συμμετέχουν στην καταπίεση των Τατάρων ή είναι μόνο τα σώματα ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πάσκου, ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η ειναι μονο τα σωματα ασφαλειας ευχαριστω πολυ κυριε πασκου ευχαριστω πολυ πολυ ενδιαφερουσα η συζητηση Πρέπει να ενημερώσω τους προσκεκλημένους μας ότι είμαι εισηγητής ε, μιας έκθεσης που ασχολείται με τη στρατιωτική κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, ιδιαίτερα μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας. Κατά συνέπεια μας ενδιαφέρει το θέμα. Θέλουμε να εντείνουμε την ευαισθητοποίηση περί της ε, στρατιωτική σπουδαιότητα αυτή τη παράνομη προσάρτηση. Γνωρίζω τώρα ότι ποια είναι η κατάσταση των Τατάρων στην Κρυμαία, αλλά και ποια είναι η κατάσταση του τοπικού πληθυσμού. Μα ενδιαφέρουν και οι δύο αυτοί οι πληθυσμοί και θέλουμε να συνεχιστεί Για να ενασχόλησή μας με το θέμα. Θα ήθελα να μάθω κατά πόσο η Ρωσία θα δημιουργήσει κάποια χερσαία οδό ε, προμηθειών προς την Κρυμαία ε, γιατί τη χρειάζεται η Κρυμαία. Ε, αν χρειάζεται κανείς να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Κρυμαία πρέπει να το μεταφέρει από τη θάλασσα ή αεροπορικός. Δεν υπάρχει τέτοιος διάδρομος. Θέλω λοιπόν να δω ποιες είναι οι προσπάθειες δημιουργίας ενός τέτοιου διαδρόμου Ταυτόχρονα, αν έχει προχωρήσει η κατασκευή αυτού του διαδρόμου προς την Κρεμαία, θα ήθελα να δω αν υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιου διαδρόμου από την Κρυμαία προς την υπερδριστερία. Ε, κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, ότι ο κύριος Πάσκου είναι ο εισηγητής μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκπονεί μια έκθεση περί της στρατηγικής κατάστασης και της στρατηγικής κατάστασης στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αναφέρεται επίση και στην παρανομή προσάρτηση τη κρυμαια Mm -hmm. Κύριε Τάνα, και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίζουμε θερμά τον κύριο Τσουμπάροφ, τον οποίο γνωρίζουμε εδώ και χρόνια. Όταν βρισκόμαστε στο Κίεβο για τη διασκέψη της Γιάλτας, έθιξα αυτό το ζήτημα, κύριε Τσουμπάροφ, που θέλω να ξαναθίξω εδώ. Ε, ανέκαθεν υπήρξε φίλο της Αρμενίας και η Τουρκία ανέκαθεν δικαιολογεί, αιτιολογεί τα κλειστά σύνορα με την Αρμενία λόγω της ε, φιλικής της σχέσης με το Αζερβαϊτζάν. Και αντιλαμβάνομαι και την αλληλεγγύη της Τουρκίας στο Ερδογάν με τους της Κρυμαία, ε, αλλά όταν ο Ερδογάν ε, επισκέφτηκε την Ουκρανία σε μια σύνδεξη τύπου με τον Ποροσέγκο υποσχέθηκε αρρωγή προς την Ουκρανία. Σίγουρα δεν θέλει να τσακωθεί με τη Ρωσία γιατί τώρα ε, διαπραγματεύεται με τον Πούτιν ε, για ε, τους αγωγούς προς τη Μαύρη Θάλασσα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Κάνει η Τουρκία περισσότερα για να βοηθήσει την κοινότητά σας γιατί ιστορικά φυσικά έχετε πολλές συνδέσεις. Γιατί όταν αρχικά είχα υποβάλει την ερώτηση μου είχατε πει ότι η Τουρκία δεν κάνει αρκετά. Επίσης κάτι άλλο. Το Μάρτιο πέρυσι είδαμε στον τύπο να έχουν ε, ζωγραφιστεί σφάστηκες πάνω στη μοναδική συναγωγή της ε, Χερσονήσου. Ε, όπως φαίνεται κάποιες δυνάμεις κατοχής ή κάποια ακραία στοιχεία ήταν υπεύθυνοι για αυτές τις βαστικές. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με τη μικρή εβραϊκή κοινότητα της Κρυμαίας, η Κρυμτσάκ και η Καράιτ, που αριθμούν μερικές χιλιάδες. Δεν έχουμε ακούσει και πολλά για αυτές τις κοινότητες το τελευταίο, το τελευταίο έτος. Αλλά σίγουρα και αυτοί θα υφίστανται διώξεις. Ευχαριστούμε. Ο κ. Οστροβίτσιος. Ευχαριστώ. Εκτιμάμε ιδιαίτερα την πρωτοβουλία Τη επιτροπή ΕΔΕ να οργανώσει αυτή την ακρόαση, τη συνάντηση σήμερα με τον κύριο Τσουμπαρόφ και τον Ουκρανό πρέσβη. Κύριε Τσουμπαρόφ, πράγματι με εξέπληξε όταν είδα τι σκηνέ από τη ρωσική τηλεόραση ο, με το κάψιμο ουκρανικών βιβλίων σαν να ήταν ε, όπλα αυτά τα βιβλία κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κλασικό παράδειγμα σκληρότητας και απολύτης της προσέγγισης της Ρωσικής ε, Ομοσπονδίας ε, όπως τη βλέπουμε μετά από την προσαρτησία της Κρυμαίας. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια σας όσον αφορά τις δραστηριότητες των Μετλής. Ποια είναι η κατάσταση. Συνεχίζονται κάποιες δραστηριότητες. Επιπλέον μπορείτε να σχολιάσετε την πιθανή στρατολόγηση των Τατάρων της Κρυμαίας ε, στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Έχουν γίνει τέτοιες ε, προσπάθειες να στρατολογηθούν ε, νέοι άνδρες από τους Τατάρους στις δύναμεις κατοχής της Ρωσίας. Και τέλος, δεν βλέπετε κάποια απειλή, κάποιο κίνδυνο για δεύτερη απέλαση των τετάρων της Κρυμαίας από την πατρίδα τους προς οπουδήποτε, προς Σιβηρία, οπουδήποτε αλλού. Ευχαριστώ για να κλείσει ο γύρος των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Σαφχάουζα. Ε, ναι κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Η ιστορία μας δείχνει ότι Ποτέ τα πράγματα δεν είναι απλά. Στην Κρυμαία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση. Όπως η συμμαχία παρενέβη ε, στη Λιβύη και στο Ιράκ, ε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη, περίπλοκη κατάσταση. Διότι, ναι, αφενός προσαρτήθηκε η Κρυμαία με ένα διάταγμα και έχουμε την αρχή βραβείας των συνόρων και μετά από το πραξικόπημα το οποίο δικαίως ονομάζω πραξικόπημα και θα σας εξηγήσω πώς ε, προετοιμάστηκε του Φεβρουαρίου 2014 βρεθήκαμε ενώπιον μια κατάσταση ε, κάπω ιδιαίτερη. Σε αυτό η Ρωσία απάντησε έχουμε μια γεωπολιτική ένταση λόγω της κατάστασης στην Κρυμαία και ενός δημοψηφίσματος όπου με μεγάλη πλειοψηφία ο λαός αποφάσισε να προσαρτηθεί στη Ρωσία. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα είχαμε φτάσει εδώ εάν είχαμε τηρήσει τις υποσχέσεις ε, που είχαν γίνει για τη μη διεύρυνση ε, στο ΝΑΤΟ ε, και τη σφαίρας επιρροής ΙΠΑ και Ρωσίας. Η συμφωνία αυτή δεν υπήρξε ποτέ θα λέει Κανεί υπήρξε αυτή η συμφωνία έχω μάρτυρε. Ε, είχα συζητήσει με τη συνάδελφό σα την κυρία και κύριε Μαζοβιέτσικη είχα την ευκαιρία να συζητήσω με την κυρία Μαζοβιέτσικη υπήρξα μάρτυρα όλων αυτών ζητώ συγγνώμη γιατί εγώ αντίθετα μέσα σε ε, πολέμησα τους κομμουνιστές και το σοβιετικό σύστημα ήμουν εκεί και πολλοί μπορούν να σα το αποδείξουν. 300 επαναστάτες ήρθαν να με συγχαρούν όταν έπεσε ο τείχο στο Στρασβούργο, εκ των οποίων ο πρόεδρος της Ουγγρική Δημοκρατίας, ο κ. Βαλέσα. Οπότε μην μιλάτε άλλο, κύριε συνάδελφε. Ε, κύριε Σεφάζερ, να σας ζητήσω να χαμηλώσετε τους τόνους. Μην προσβάλλετε τα μέλη, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, έχετε δίκιο, αλλά όταν μου επιτίθενται υποχρεωμένο να απαντήσω. Στην πολύπλοκη κατάσταση αυτή λοιπόν πρέπει να βρούμε μια λύση. Έχουμε πρώτα απ' όλα τι συμφωνίε του Μίνσκ, πρέπει να προσπαθήσουμε να μπούμε σε μια ειρηνευτική διαδικασία, σε μια διαδικασία διαλόγου. Είμαι πεπισμένο ότι θα καταφέρουμε να βρούμε λύσει. Πρέπει να πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή στην Ουκρανία οι επαναλαμβανόμενε αυτοκτονίες των ε, μέλων της αντιπολίτευσης από ό,τι φαίνεται είναι συλλογικέ ε, ε, στην Ουκρανία. Υπάρχει η φτώχεια, η χρεοκοπία, απουσία μεταρρυθμίσεων. Μόνο 6% υποστήριξη έχει η τρέχουσα κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν ένα βαθύ πρόβλημα το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί μόνο με διάλογο και διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό υποστηρίζω πλήρως τις συμφωνίες του Μίνσκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στέτινα παρακαλώ. Please, colleagues. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Ο κύριος Στέτινα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κάτι πολύ σύντομο από πλευρά μου, μετά από αυτά που είπε ο κύριος Σαφχόιζα. Ο κύριος Σαφχόιζερ είναι το ιδανικό παράδειγμα για το τι επιχειρήματα χρησιμοποιεί κανείς όταν δεν έχει περάσει όσα περάσαμε εμείς που ήμασταν στο πρώην ε, Σοβιετικό στρατόπεδο. Ξέρουμε τι σημαίνει κατοχή από Σοβιετικό στρατό. Και τώρα ορισμένοι διαπιστώνουν τι σημαίνει να κατέχεσαι από Ρωσικό στρατό. Αυτά για αυτά που είπε ο κύριος Σαφχόιζα. Για τον κύριο Τσουμπάροφ και τον ε, κύριο Πρέσβη θέλω να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην ε, αντιπροσωπεία μας που επισκέφθηκε την Αρμενία το Ερεβάν για την ετήσια συνεδρίαση του Euronest. Είναι μια κοινοβουλευτική συνέλευση των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας. Και την προηγούμενη λοιπόν εβδομάδα εγκρίναμε ένα πολύ κατηγορηματικό ψήφισμα για την προσάρτηση της Κρυμαίας. Και ήμασταν πολύ σαφείς. Όσο για τις κυρώσεις. Τονίσαμε ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την Κρυμαία όταν συζητάμε για τις κυρώσεις. Αυτά που είπατε είναι πολύ σωστά. Όσο η Κρυμαία παραμένει υποκατοχή, δεν μπορούν να αρθούν οι κυρώσεις. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω. Στη χώρα μου, την Τσεχία, την επόμενη εβδομάδα θα παρευρεθούν Αμερικανοί στρατιώτες που φεύγουν από τις βαλτικέ χώρες και μετά θα περάσουν από την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία για να επανέλθουν στις βάσεις τους ε, στη Γερμανία. Είναι μία απόδειξη ότι είμαστε προπαρασκευασμένοι από στρατιωτική πλευρά. Έχουμε το αναγκαίο επίπεδο ετοιμότητας και είναι και μία επίδειξη δύναμης στα πλαίσια αυτά. Θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο Τσουμπάροφ τον πρόεδρο των Τατάρων της Κρυμαίας. Δεν θα έπρεπε επιτέλους να δείξουμε και το επίπεδο ετοιμότητάς μας από στρατιωτική πλευρά στην περιοχή της ε, Μαύρης Θάλασσας και στο έδαφος της Ουκρανίας. Ευχαριστώ πολύ. Τι άποψη έχετε από αυτού. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Τούνε Κέλλα. our Ukrainian and Tatar friends. And... Ευχαριστώ. Καλωσορίζω τους φίλους μας από τους Τατάρους της Κρυμαίας και να επενθυμίσω ότι αυτά τα είδαμε και στις βαλτικές χώρες το 1940 και το γεγονός ότι δεν αναγνωρίστηκαν οι προσαρτήσεις που έγιναν τότε από τη Ρωσία από, τα δημοκρατικά χώρα, από, τις δημοκρατικές χώρες ότι παρά τις τρομερές πιέσεις της Real Politik για 50 χρόνια δεν αναγνωρίστηκαν αυτές οι προσαρτήσεις των βαλτικών χωρών, αλλά τελικά επανήλθαν στην κατάσταση ανεξαρτησίας. Άρα πρέπει να εμείνουμε στην πολιτική μη αναγνώριση της προσάρτησης της Κρυμαίας. Και όπως υπόθηκε, δεν θα πρέπει να εκτραπούμε από άλλα γεγονότα. Γιατί μπορεί να επιδιωχθεί η εξομάλυνση Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί για να αρχίσουμε συζητήσεις, για να μειωθούν οι κυρώσεις, για παράδειγμα. Η θέση μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να εμείνουμε στις κυρώσεις μέχρι ότου να υπάρξουν σαφή δείγματα ότι θα ακυρωθεί η προσάρτηση και θα αποκατασταθεί η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ανησυχώ για αυτά που είπατε για τις έρευνες που κάνει η FSB, η μυστική ρωσική υπηρεσία, για τους ε, διαδηλωτές υπέρ της Ουκρανικής εδαφικής ακεραιότητας. Και το μήνυμά μου προς τον ε, κύριο Πρέσβη, ή μάλλον η ερώτησή μου, είναι θεωρείτε ότι σε αυτή τη φάση η Ουκρανία χρειάζεται δυτική στρατιωτική βοήθεια, δηλαδή αμυντικά όπλα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες ρωσικές επιθέσεις. Δεν είναι αναγκαίο επίσης να επεκταθούν περαιτέρω οι κυρώσεις. Για παράδειγμα, συμπεριλάβουν και όσους είναι υπεύθυνοι για τη ρωσική προπαγάνδα, την παραπληροφόρηση, τη δυσφήμιση άλλων κρατών και ε, λαών. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ ο κύριος Μποστινάρ. Ευχαριστώ. Εξαιρετικοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές, διότι η αποτίμηση που έκαναν για την κατάσταση στην Κρυμαία δείχνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με τη ρωσική προπαγάνδα και την πέμπτη φάλαγγα σε πολλά κράτη-μέλη και μιλώ και εδώ για κάποιους εκπροσώπους τους εδώ, στο Κοινοβούλιο. Αυτά που ακούσαμε από αυτούς δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πολιτική σχεδιάστηκε με απόλυτη ακρίβεια από τη Μόσχα και από τον Πούτιν και ε, εξάλλου ε, υπήρξε στο μεταξύ, έγινε στο μεταξύ και η περίφημη συνέλευση του Πούτιν όπου μας εξήγησε ακριβώς πώς και τι έκανε και γιατί το έκανε και έρχονται στην και να, να μας αποδείξουν τι την, ότι είναι, λειτουργεί καλή την πίστη ο Πούτιν το Φεβρουάριο όταν αποφάσισε την κατοχή της Κρυμαίας ο Πούτιν, όταν δεν υπήρχε καμία αξίωση σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και επιθέσεις κατά των ρωσόφωνων της Κρυμαίας, τίποτα τέτοιο δεν υπήρχε, ήταν μόνο μία υπερελιστική απόπειρα της Ρωσίας που εφαρμόστηκε με το στρατό χωρίς διακριτικά σήματα. δική του ήταν οι στρατιώτες. Αυτή είναι η πραγματική ε, ιστορία και μας την επιβεβαιώνουν οι προσκεκλημένοι μας. Δεύτερη παρατήρηση, η εθνική καθαρση όπως μας την περιγράψατε σήμερα. Τι μας δείχνει ότι αυτοί που υφίστανται την καταστολή, αυτοί που ε, έχουν επεμπολίσει τα ε, νόμιμα δικαιώματά του, γιατί δεν πρόκειται μόνο για τους Τατάρους, αλλά για όλους όσους πλήττονται από την ρωσική κατοχή. Μα ε, έρχεστε και ισχυρίζεται η Ρωσία ότι προστατεύει τους ρωσόφωνους. Είναι απαράδεκτο επιχείρημα και παραβιάζει οποιαδήποτε έννοια διεθνούς δικαίου, οποιοδήποτε πρότυπο Συμβουλίου της Ευρώπης ή ο ΑΣΕ. Υπάρχει σαφώς αντίφαση ανάμεσα στη ρωσική προπαγάνδα και τις ιστορίες της πέμπτης φάλαγγας σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης από πλευράς ε, θεσμοθετημένων πολιτικών κομμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πραγματικότητας. Παρακαλώ, ας μην συνεχίσουμε με την έλλειψη αποφασιστικότητας να πάυσει αυτή η χρηματοδότηση. Ε, θα Πρότεινα μάλιστα να θεσπιστεί ένας μηχανισμός ούτως ώστε όσα πολιτικά κόμματα αντιμάχονται τα συνταγματικά πρότυπα και τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτόματα να διαγράφονται από τα Μητρώα διότι είναι άμεση απειλή προς την εσωτερική ασφάλεια όλων των κρατών με της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά που έγιναν στην Κρυμαία, το, μας το επιβεβαιώσατε κι εσείς, η Κρυμαία τι έχει γίνει ε, στην Κρυμαία, ότι με το πρόσχημα της προστασίας των ρωσοφόνων η Ρωσική Ομοσπονδία μετέτρεψε την Χερσόνησο της Κρυμαίας στην ισχυρότερη στρατιωτική βάση αυτή τη στιγμή στον έξινο Πόντο και το πρόβλημα είναι ότι απειλείται όχι μόνο η σταθερότητα της Μαύρης Τάλασσας αλλά και της ευρύτερης περιοχής ε, διότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή βρίσκεται είναι αναγκασμένο να ε, χρησιμοποιήσει ε, το δυναμικό που έχει για να αντιμετωπίσει τις καθημερινές πλέον προκλήσεις και παραβιάσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από αυτήν την στρατιωτική βάση θυμάστε την συμφωνία της, ε, του Μονάχου, είχαμε το, τον Πετέν, το, τον Τσάμπερλεν, τι κάναμε εμείς, ε, ακολουθήσαμε την γραμμή Τζαλαδιέ, τη γραμμή Πεντέν Τσάμπερλεν, τι κάναμε, αποτρέψαμε τον πόλεμο, μήπως αποτρέψαμε έτσι ε, τον Χίτλερ και τον αναγκάσαμε να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, καμία σχέση. Θα έλεγα λοιπόν ότι Καλύτερο θα ήταν να αφήσουμε τις ψευδεστήσεις και την ουτοπία σε σχέση με την αποδυνάμωση των κυρώσεων ε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, χάρη στο Συμβούλιο, μπορέσαμε να διατηρήσουμε τις κυρώσεις και πέραν αυτό να συνεργαστούμε στενότατα με τον ΝΑΤΟ, διότι σε με αυτές τις τραγικές εξελίξεις η μοναδική άμυνα που έχουν οι χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης ε, είναι η προστασία του ΝΑΤΟ. Ωραία και τα λόγια, αλλά δεν είναι αποτελεσματικά κατά του ε, ε, πυροβολικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ. Thank you, colleague. Now... Ευχαριστούμε κύριε συναδέλφε, κύριε Σμαζουλίτσο. Dziękuję bardzo, Madam e, President. Ladies and gentlemen, first of all, uh, thank you very much for inviting uh, our friends from uh, Crimea. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε που προσκαλέσατε τους φίλους μας, τους εκπροσώπους των Λιτατών της Κρυμίας. Not a very sensitive situation, but a very difficult situation, considering... Βρισκόμαστε ενώπιον μια κατάσταση ε, που παραβιάζει το διεθνέ δίκαιο όλε τι συμφωνίε το πλαίσιο όλων των συμφωνιών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειδικότερα μετά από την κατοχή της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Μετά από τα γεγονότα στην Ανατολική Ουκρανία, τον πόλεμο εκεί όπου η Ρωσία και οι αυτονομιστές ε, προσπάθησαν να καταλάβουν περισσότερη γη, ο κόσμος τώρα αρχίζει να ξεχνάει την Κρυμαία και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εξαγωγή αυτή εδώ τη συνάντηση και των επόμενων τέτοιων συναντήσεων. Γιατί ξέρετε, μιλάμε για χαλάρωση των κυρώσεων προ τη Ρωσία ή τη λήξη των κυρώσεων σε περίπτωση που η Ρωσία συμμορφωθεί με τη συμφωνία του Μίνσκα. Αλλά οποιαδήποτε συμφωνία θα κάνουμε θα πρέπει να σχετίζεται με την κατάσταση στην Κρυμαία, να επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση. Μην ξεχνάμε την Κρυμαία η Κρυμαία πρέπει να παραμένει κεντρικό θέμα στην προσέγγιση μας της κατάστασης στην Ουκρανία διότι κυρίες και κύριοι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ρωσία κινείται πολύ έξυπνα αν αύριο γίνει κάτι καινούριο σε κάποιο άλλο κομμάτι της Ουκρανικής επικράτειας ή αν συμβεί κάτι νέο όπως η Ρωσία να προσπαθήσει να ε, αμφισβητήσει τα σύνορα ενός ευρωπαϊκού κράτους πιθανότατα θα ξεχάσουμε αμέσως την Ανατολική Ουκρανία και θα πάψουμε να μιλάμε για την Κρυμαία. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τα ζητήματα αυτά. Οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να σχετίζεται με την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Είναι πολύ σημαντικό. Διότι όπως βλέπετε πολλοί Ευρωπαίοι και άλλοι πολιτικοί λένε ότι η ρεαλιστική πολιτική θα πρέπει να ξεχάσει την Κρυμαία. Η Κρυμαία έχει χαθεί. Αυτό δεν αληθεύει. Δεν πρέπει να πάψουμε να έχουμε στο κέντρο της σκέψης μας την εδαφική κυριαρχία ενός ευρωπαϊκού κράτους και την Κρυμαία. Διότι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας τώρα είναι μια εντελώ διαφορετική κατάσταση. Παραβιάζει τις αρχές μας, τις αξίες μας, τη δημοκρατία μας. Έχουμε περάσει σε ένα καινούριο κόσμο. Όλοι μαζί πρέπει να πολεμήσουμε σε αυτό τον καινούριο κόσμο. Διότι αλλιώς πραγματικά στο μέλλον θα γίνει πραγματικός πόλεμος. Θα πάψουμε να χρησιμοποιούμε ήπια μέτρα. Κυρίες και κύριοι, να κάνω ξανά έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμά ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να εκπονήσουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν έχουμε καμία ακόμα πραγματική στρατηγική, ούτε πραγματικά μέτρα και ταυτόχρονα πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα με τους φίλους μας ε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και άλλες δημοκρατικές χώρες ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Διαφορετικά δεν θα σταματήσει να επιδεινώνεται στο μέλλον. Ευχαριστούμε, αξιότιμοι συνάδελφα. Έχουμε πλέον ελάχιστο χρόνο. Να ζητήσω στα μέλη του πάνελ, ε, ξεκινώντας από τον αξιότιμο πρέσβη κύριο Ηλισίευ και μετά τον κύριο Τσουμπάροφ, ε, ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις και να σχολιάσουν περαιτέρω. Δυστυχώς έχουμε ελάχιστο χρόνο. Παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φατίγκα. Εν συντομία, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη που εκφράζεται με την Ουκρανία επί αυτού του πολύ σημαντικού θέματος. Να σας διαβεβαιώσω ότι οι Ουκρανικές αρχές, ο πρόεδρος, η κυβέρνηση της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται ώστε να πάρουν πίσω ε, την Κρυμαία. Αγαπητοί φίλοι, για να είμαστε δίκαιοι, αυτά παρουσίασε μόλις ο κύριος Τσουμπάροφ. Δεν είναι παρακομμάτι της συνολικής εικόνας ε, των όλων των πιθανών παραβιάσεων, των παραβιάσεων ανθρωπιστικών διεθνών προτύπων και αρχών υπογράμμισε την κατάσταση ο κ. Σουμπαρόφ των Τατάρων της Κρυμαίας αλλά όπως υπόθηκε εδώ η κατάσταση είναι ολόενα επιδεινούμενη και όσον αφορά άλλες ε, μειονότητες γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στην Κρυμαία δεν έχουμε μόνο ρωσόφωνους αλλά και εβραϊκή μειονότητα οι οποίοι απλά έφυγαν διότι οι συνθήκες διαβίωσης εκεί είναι επικίνδυνες, ε, καταστολή καθημερινά, παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό απλά έφυγαν. Ίδια κατάσταση και για τους Ουκρανούς. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γη μας. Έχουν κλείσει βιβλιοθήκες, ε, απαγορεύονται τα ουκρανικά βιβλία. Μην ξεχνάμε και την κατάσταση όσον αφορά την Ουκρανική Εκκλησία. Γι' αυτό έχουμε εδώ τους εκπροσώπους της ε, Ουκρανικής Εκκλησίας ε, διότι και για αυτούς η κατάσταση είναι τρομακτική. Υπάρχει πλήρης παραβίαση των θρησκευτικών δικαιωμάτων ε, των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και θα πρέπει να εκφράσει, να απασχολήσει την παρούσα επιτροπή είναι στρατιωτικοποίηση της Κρυμαίας. Θα έλεγα μάλιστα η ύπαρξη πυρηνικών όπλων στην Κρυμαία. Είναι κάτι που επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε να συζητήσουμε, διότι η τοποθέτηση πυρηνικών κεφαλών όχι μόνο θα παραβιάσει όλους ε, τους διεθνείς νόμους και τις αρχές, αλλά όπως σημειώθηκε θα αποτελέσει τεράστια απειλή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής, καθώς και ολόκληρης της Ευρώπης. Επίσης, αγαπητοί φίλοι, ακούσαμε μια ερώτηση όσον αφορά τα αμυντικά οπλικά συστήματα, κατά πόσο η Ουκρανία τα χρειάζεται ή όχι. Ναι, πράγματι, χρειαζόμαστε αμυντικά συστήματα για να υπερασπίσουμε την Ουκρανία σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χαρτί των Ηνωμένων Εθνών, το δικαίωμα ε, για άμυνα. Αλλά πρέπει να υπερασπίσουμε όχι μόνο τους στρατιώτες μας, Πρέπει να υπερασπίσουμε και τους αμαχούς πολίτες μας. Χρειαζόμαστε αυτά τα όπλα για να αποτρέψουμε τον εισβολέα. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι στον τομέα αυτό έχουμε επιτύχει κάποια σημαντική πρόοδο μέχρι στιγμής. Όπως καταλαβαίνετε για πολλές αιτίε δεν μπορώ να σας περιγράψω το θέμα αυτό λεπτομερώς, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και όπως φαντάζεστε υπάρχει πολλοί κόσμος που θα ήθελε όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις ε, ε, συμβάσεις. Ε, είμαστε ευγνώμονες σε κάποια κράτη-μέλη που μας βοήθησαν και είμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι με την ενίσχυση οι στρατιωτικές μας δυνάμεις θα ενισχυθούν όλο και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ισχυρές ε, που ελπίζουμε να γίνουν ισχυρότερα στην Ευρώπη με τη δική σας βοήθεια, με τη δική σας αλληλεγγύη. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε πρώτα απ' όλα να αντισταθούμε στο Ρώσο εισβολέα στην περιοχή του Νταμπάσα και να ξαναπάρουμε την Κρυμαία. Και για να κλείσουμε ε, λίγο πιο, σε μια πιο θετική νότα, αγαπητοί φίλοι, θα κάποια στιγμή οι ρωσικές αρχές και ο ρωσικός λαός και ο κύριος Αφάζεν μάλλον θα ζητήσουν συγνώμη για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κρυμαία. Όσο τον ε, συντομότερο τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κ. Τσουμπάροφ. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομο γιατί κατάλαβα ότι δεν υπάρχει χρόνο. Ε, με συγχωρείτε αν θα μπορέσω να απαντήσω όλε τι ερωτήσει. Κύριε Γκάλερ, αναφερθήκατε στην στρατιωτικοποίηση ορισμένων περιοχών. Δεν είμαι η για αυτά τα θέματα, αλλά είναι σαφές ότι η Κρυμαία στρατιωτικοποιείται με ταχύ ρυθμό και κυρίως το Τσανκούι και το Κασπερικό στο βορρά. Εκεί έχουν στρατοπεδέψει πολλά στρατεύματα. Είναι περιοχές που είναι επίση κοντά στη θάλασσα. Και έχουν εγκατασταθεί ε, τελευταίας λέξεις ε, πυραυλικά συστήματα σε αυτές τις περιοχές. Για τις ερωτήσεις του κυρίου Πάσκου. Βεβαίως, μέσω θαλασσίας οδού μπορούν να μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτό αρκεί για τους Ρώσους. Αλλά βέβαια για να μπορέσει και ο πληθυσμός να πάρει ε, τις αναγκαίες προμήθειες, όλα όσα χρειάζεται, χρειάζεται χερσαίος διάδρομος. Θα κάνουν ε, αυτό που χρειάζονται για να αποκτήσουν αυτόν τον χερσαίο διάδρομο. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που δεν μπορώ να αποτιμήσω, αλλά η απειλή είναι σαφής για τις ερωτήσεις από τον πολύ καλό φίλο μου τον κύριο Τάνοκ. Το συζητάμε αυτό που είπατε συνεχώς και προσπαθούμε να επηρεάσουμε την κατάσταση. Πριν από μερικές μέρες ε, ο κύριος Τζαμίλεφ και εγώ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχαμε μια διεξοδική συζήτηση με τον κύριο Ερντοάν. Είναι το θέμα των σχέσεών μας με την Τουρκία και πόση βοήθεια μας δίνει. Και ελπίζω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ γιατί η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ελπίζω ότι θα βρούμε το σωστό τρόπο να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για την ε, εβραϊκή κοινότητα στην Ουκρανία. Το ανέφερε και ο κύριος Πρέσβης. Ναι. Ε, έχουν μεταναστεύσει πολύ. Αυτό είναι σαφές. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους Ρώσους αλλά και άλλες μειονότητες. Ως ε, τάταροι της Κρυμαίας, όπως ξέρετε, εκτοπιστήκαμε από τη χώρα μας για 50 χρόνια και μόλις επανήλθαμε. Καλούμε λοιπόν όλους τους τατάρους να μείνουν στα εδάφη τους, ανεξάρτητα από αυτά που υφίστανται. Για το θέμα του πώς λειτουργεί η νομοθετική μας συνέλευση, το Μετζλής. Συνεδριάσαμε προχτές, μέσω Skype, διότι οκτώ μέλη μας ζουν ε, στην ε, υπηρετική Ουκρανία. Οι υπόλοιποι είναι στην Κρυμαία. Αλλά η κατάσταση βέβαια είναι πολύ δύσκολη σε σχέση με το παρελθόν. Από ό,τι φαίνεται, οι προθέσεις ε, των αρχών κατοχής είναι να αλλάξουν το, το Μετζλής ούτως ώστε να μπορέσουν να το έχουν υποχείριό τους. ούτω ώστε να βγαίνει το Μεσλή να λέει ότι εμείς εγκρίνουμε αυτήν την ε, κατοχή. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Μετά τον Απρίλιο του 2014 δεν αποκλείουμε οποιαδήποτε ενέργεια. Θα μπορούσαν να εκτοπίσουν και πάλι ολόκληρες κοινότητε, ολόκληρα έθνη. Κρίμα που έφυγε ο κύριο Σαφχάουζερ. Είναι η δεύτερη φορά που ακούω αυτά που λέει. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ πλήρω με ε, ένα θέμα Ίσως θα μπορούσε κάποιος να τον ενημερώσει. Πρέπει να μιλήσουμε για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Είμαστε μία εθνότητα, η Τάταρη της Κρυμαίας. Μία εγχώρια εθνότητα. Δεν λέμε ότι θα έπρεπε να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης σε οποιαδήποτε ομάδα πληθυσμού, οπουδήποτε, ορισμένες φορές ε, λέει ε, σωστά και μετά όμως κάνει το αντίθετο ακριβώς όπως ο Πούτιν. Με συγχωρείτε πρέπει να το πω. Βεβαίω είπε ότι δεν τηρήθηκε η υπόσχεση για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αλλά πείτε μου, ποιος ε, τήρησε τη συμφωνία της Βουδαπέστης, η Ρωσία. Κρίμα που δεν είναι παρόν ο κύριος Σαφχάουζ να με ακούσει. Για την ερώτηση του κυρίου Στέτινα. Βεβαίως, ε, σε ευχαριστώ πολύ που το επιβεβαιώσατε ότι κανείς δεν μας ξεχνά. Ίσως να μην ε, ήμουν απόλυτα αντικειμενικός όταν είπα ότι όλοι μας ξεχνούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτά που λέτε και για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων στην Νότια Ουκρανία. Το είπε και ο κύριος Πρέσβης. Χρειαζόμαστε όπλα ακριβίας. Αυτό είναι σαφές. Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις, ιδιαίτερα στο νότο της χώρας μου, πρέπει να λάβουν σύγχρονο εξοπλισμό. Και το ερώτημα του κυρίου Κέλαμ. πρέπει να μας δώσετε στρατιωτικό εξοπλισμό ή να επιβάλλετε κυρώσει και τα δύο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, να εξυγχρονίσουμε τη χώρα μας, να προωθήσουμε τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ κύριε Μποστινάρου για τα σχόλιά σας με τα οποία συμφωνώ απόλυτα. Και για τον κύριο Φοντουλίτσα επίσης τον ευχαριστώ για το πώς πολύ σωστά θέσατε τα θέματα. Κρίμα που έφυγε ο διπλανός σας, ο κύριος Σαφχάουζερ, γιατί ασχοληθήκατε και με αυτά που είπε. Αλλά δεν σας άκουσε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής μας και άλλων Επιτροπών. ε, αξιοπρεπείς, συγγνώμη, διακεκριμένοι εκπρόσωποι από πλευράς όλων των συναδέλφων μου, την κυρία Μπρούνοβα και τον Αρχιεπίσκοπο Κλίμεντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω ε, η κατάσταση να βελτιωθεί ούτως ώστε όλος ο λαός της Κρυμαίας να δει ότι παίρνει έμπρακτη βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη, κύριε Τσουμπάροφ για αυτήν την ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Κυρίες και κύριοι, αν ε, μου επιτρέπετε, να δώσω τώρα για πολύ λίγο το λόγο στον Αρχιεπίσκοπο Κλίμεντα της Κρυμαίας. Συμφωνείτε? Ωραία. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, και Πρέσβη, με τιμά ιδιαίτερα η σημερινή πρόσκληση για να μετάσχω στη συζήτηση για την Κρυμαία. Έχει περάσει ένας χρόνος από την προσάρτηση, ένας πολύ δύσκολος χρόνος και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συζητάτε για προβλήματα που είναι πραγματικά. Δεν δεν υπάρχει καμία υπερβολή σε αυτή την αξιολόγηση που ακούσατε. Χρειαζόμαστε ε, στρατιωτική υποστηρίξη ώστε να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε την εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Χρειαζόμαστε βοήθεια επίσης για τις κυρώσεις. Γιατί? Διότι οι κυρώσεις επηρεάζουν πραγματικά τις εξελίξεις, τις πολιτικές εξελίξεις. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας ώστε να επιστρέψει η Κρυμαία στην επικράτεια της Ουκρανίας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό είναι ένα θέμα ασφαλείας και για την ευρωπαϊκή κοινότητα σήμερα μετατρέπεται σε μία πελώρια στρατιωτική βάση η χερσόνησος της Κρυμαίας. Και η στρατιωτική ικανότητα υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε συνθήκη έχει υπογραφεί με τη Ρωσία. Είναι καταστροφικές οι εξελίξεις για την Ουκρανία. Παραβιάζεται η Ουκρανική νομοθεσία, τα σύμβολα της Ουκρανίας, τα εθνικά σύμβολα της Ουκρανίας πλέον καταδικάζονται μέσω του νόμου ε, κατά των εξτρεμιστών. Ένα 16χρονο παιδί ξυλοκοπήθηκε ε, μέχρι θανάτου μόνο και μόνο επειδή μίλησε ουκρανικά. Υπάρχουν άπειρες παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθημερινά και θα ήθελα να απευθύνω μια θερμή έκκληση να μην Λυσμονείτε το θέμα της Ουκρανίας, αλλά να εγγράφετε το σημείο ε, στην μερήση διάταξη όλων των συζητήσεων. Σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετάσχω στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Αρχιεπίσκοπε Κλίμεθ. το Κλίμεθ. Και θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο σε συνεργασία με την Επιτροπή ΑΦΕΤ ε, για την κοινή αποστολή Σέντε και ε, που έγινε στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Debriefing για την ε, αποστολή της ε, υποεπιτροπής μας στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα. δύο ημέρες περίπου, λίγο περισσότερο από δύο δύο διήρκησε η αποστολή και είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με όλους τους σημαντικούς συνομιλητές σε πολιτικό επίπεδο και επίπεδο κοινωνίας των πολιτών στην Ουκρανία εκτός από τον πρόεδρο Ποροσέγκο αλλά ήταν πολύ στενά τα χρονικά όρια που είχαμε οι Ουκρανικές αρχές Επίσης, ε, εργάζονταν και για την Σύνοδο Κορυφής. Ε, παρόλα αυτά, μπορέσαμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Ο κύριος Κλίμκιν, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, και η κυρία Γκαριμπαλέγκοφ, η πρώτη αναπληρώτρια που ήταν ε, η ομόλογός μας σε πάρα πολλές συνεδριάσεις έδειξε υποδειγματικό επαγγελματισμό και μας ενημέρωσε για την κατάσταση. Μας ενημέρωσαν επίσης για το αίτημα της Ουκρανίας που υπέβαλε στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων ώστε να υλοποιηθεί σωστά η Συμφωνία του Μίνσκ. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή Άμυνας ε, θα είναι συναρμόδιες για την απόφαση αυτή. Πρέπει λοιπόν να προβούμε σε μια αξιολόγηση τη κατάστασης. Επίσης, παραβρεθήκαμε στα εγγένεια του κτηρίου της νέας ε, Συμβουλευτικής Αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο κέντρο του Κιέβου απέναντι από το Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Εξωτερικών και Δικαιοσύνης στη συνέχεια την επόμενη μέρα συνεργασία με του συναδέλφου από την Επιτροπή Προπολογισμών έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τη χρηματοδότηση των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης μετά από την αποστολή της EUAM, αυτής της συμβουλευτικής αποστολής. Στη συνέχεια συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Αμήνης και το επιτελείο του. Ήτανε πολύ καλή και ειλικρινή η ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, στη Χόβνεράντα στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ε, γινόταν τότε και μια σύσκεψη της Επιτροπής ε, Άμυνας ε, και συμμετείχαμε και εμείς. Πολλοί έχουν, είχαν δραστηριοποιηθεί νωρίτερα σε στρατιωτικές εξάλλου δράσεις περάσπιση της εδαφικής ε, ακυρότητας Ουκρανίας. Σε συνέχεια ο κύριος Τουρτσίνα, ο Γενικός ε, Γραμματέας ε, υπεύθυνο για θέματα αμήνη από, από την Προεδρία της Ουκρανίας συναντήθηκε μαζί μας. και ένα, ε, κάποιοι από εμά ε, μπόρεσαν να συναντηθούν και με τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας. Έτσι ολοκληρώθηκε εξάλλου και η αποστολή μας. Ο κύριος Γκάλλου και η κυρία Γκόμες μπόρεσαν να μεταβούν και στην Ανατολική Ουκρανία και θα ήθελαν να σας ενημερώσουν γι' αυτό. Δεν θέλω να μονοπολίσω το λόγο, κύριο Γκάλε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όπως είπαμε, μαθαίνουμε πολλά σε αυτή την επίσκεψη στην Ουκρανία αντιληφθήκαμε για άλλη μια φορά πόσο πλευρέ είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει αυτή η χώρα. Επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά την ομόφωνη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη σημερινή κρίση. Η θέση μας είναι αδιαμφισβήτητη, όπως είναι και τα όσα υποστηρίζουμε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η επίσκεψή μας έγινε παράλληλα μαζί με την ε, επίσκεψη της Επιτροπής Προπολογισμού για τους γνωστούς λόγους. Ξέρετε, χορηγούμε άμεσα και έμεσα πολλά χρήματα σε αυτή τη χώρα για να αποφευθεί χρεοκοπία, για να υπάρξει κάποια σταθεροποίηση. Και όπως πολύ σωστά είπατε, παρευρεθήκαμε στα εγγένεια της Συμβουλευτικής Επιτροπής ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει για να βοηθήσει σε νομοθετικά θέματα και σε θεσμικές αλλαγές παρέχοντας τη δική μας εμπειρογνωμοσύνη των τελευταίων 25 ετών. Η αρρωγή αυτή αφορά την νομοθεσία περί ε, δημοσίου, περί γενικού εισαγγελέα, περί ε, γραφείου καταπολέμησης της διαφθοράς. Αφορά πολλά ε, νομοθετικά πακέτα που πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Η κυβέρνηση έχει εκφράσει στο κοινοβούλιο πολιτική βούληση για αλλαγές αλλά υπάρχει μεγάλη αντίσταση οπότε πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό χρειάζονται επιδέξει χειρισμοί ε, και πολύ καλές έμπειρες συμβουλές επί τόπου ώστε να κινηθούν τα πράγματα προς την επιθυμητή οδό όταν συνέντησα με τον Πρωθυπουργό ε, καθυστέρησε στη συνέντηση διότι μόλις είχε μια συνέντηση με τον πρόεδρο και ήταν ορατά ανήσυχο, ε, διότι μόλις είχαν μάθει ότι για πρώτη φορά μετά από τη συμφωνία απόσυρσης ε, του βαρέως οπλισμού στο βόρειο μέρος στην περιοχή του Λουγκάνσκ χρησιμοποιήθηκαν ξανά πύραυλοι και βαρύ πυροβολικό και για άλλη μια φορά πιστεύω συνολικά η εκτίμηση που κάναμε εμείς είναι ότι η εκεχηρία παύση του πυρός ε, παραμένει επισφαλής. Ε, εγώ συζήτησα με την Ανακόμε, με, με, την με διάφορους εμπειρογνώμονες και αυτά που μάθαμε από τον ΟΑΣΕ είναι πόσο πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες ε, αισθάνονται παράξενα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους πυροβολισμού που έρχονται από την άλλη πλευρά. Γνωρίζουμε ότι οι Ουκρανοί πρέπει να υπακούν ε, στα όσα συμφωνήθηκαν, ε, δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας ε, και η Ρωσία, η Μόσχα λέει ότι αυτοί πρέπει να κάνουν ό,τι συμφωνήθηκε όχι εμείς. Οπότε η στρατιωτική κατάσταση είναι επισφαλής, οι εντάσει παραμένουν, ο ΑΣΕ δεν έχει πρόσβαση σε ολόκληρη την περιοχή που κατέχεται από τους ε, επαναστάτες, ε, ειδικότερα μεταξύ Μαριούπολης και τον Νοβοαγιόφσκ στα ρωσικά σύνορα. Εκεί δεν υπάρχει πρόσβαση. Εκεί όπου έχει συγκεντρωθεί ε, το μεγαλύτερο μέρος του βαρέως προβολικού. Και σε αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε εμείς πολιτικά ως μέλη του Κοινοβουλίου. Εμείς είμαστε μέλη του ΟΑΣΕ όπως είναι και η Ρωσία. Πρέπει να επιμείνουμε να δοθεί πλήρης πρόσβαση στον ΟΑΣΕ και ειδικότερα στην αποστολή παρακολούθηση στην Ουκρανία ώστε να εκτιμήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί επί τόπου και τι συμβαίνει. Φυσικά συνομιλήσαμε με διαφόρους εκπροσώπους διαφόρων ε, ε κομμάτων από το Κοινοβούλιο. Ε, όλοι γνωρίζουν, για να το πω λίγο δραματικά, ότι αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία να μεταρρυθμίσουν τη χώρα. και να σταματήσουν τον εισβολία εκεί που βρίσκεται χωρίς να προχωρήσει άλλο. Βάσει των όσων είδαμε και ακούσαμε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα με αυτή την ε, συμβουλευτική αποστολή ε, εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη γενική προσέγγιση και ειδικότερα επί των ζητημάτων του ΑΣΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει στη μεταρρύθμιση της δομής των δυνάμεων ασφαλείας. Οι αστυνομικέ δυνάμεις και οι αρμόδιοι για την εσωτερική ασφάλεια θα πρέπει να υιοθετήσουν μια εντελώς νέα δόμη ε, και πρακτική επιτόπου ώστε να εξυγχρονιστεί πλήρω η αστυνομική δύναμη. Πολλές φορές ε, ρώτησα να μάθω την ιεραρχία του τακτικού στρατού και τα διάφορα τάγματα που χρηματοδοτούνται με κάποιο τρόπο ε, μας επιβεβαίωσαν ότι είτε βρίσκονται υπό τη διοίκηση του στρατού είτε υπό τη διοίκηση του Υπουργείου Εστερικών. Αυτό μας είπαν. ότι δεν υπάρχει ε, στρατιωτική ομάδα που δεν είναι υποπολιτικό έλεγχο ε, και αλλού οι εντολές του Κιέβου δεν είναι πολύ σημαντικές για κάποια τάγματα. Υπαρμένουν ε, ερωτηματικά δηλαδή για όλο αυτό το θέμα και η κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οτιδήποτε έχουν συμφωνήσει με τη διεθνή κοινότητα μέσω του Μίνσκ να υλοποιείται και επιτόπου. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω, ε, κάτι πολύ θετικό που παρατηρήσαμε στην Ουκρανία, ότι το Συμβούλιο της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη εβδομάδα συνέδεσε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνιών του Μίνσκ με πιθανή άρση των κυρώσεων ή το αντίστροφο εφόσον για όσο καιρό δεν έχει εφαρμοστεί πλήρω το Μίνσκ, δεν πρόκειται να έρθουν κυρώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Είμαστε μια μικρή αποστολή, μόνο τέσσερα μέλη. Και ο κύριο Φρόιντ ήταν παρόν. Θα θέλατε να μας σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Δεν είμαι τόσο συναισθηματικός όσο η Άννα Γκόμες. Άρα θα είμαι αρκετά λιτός στις διατυπώσεις μου. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση μόλις φτάσαμε στο Κίεβο ήταν αυτή η τρομερή αντίθεση ότι λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα ε, ανατολικά του Κιέβου παρά την κατάπαυση του πυρός πολλοί πεθαίνουν ένα βίο θάνατο, ενώ το Κίεβο ήταν απόλυτα ειρηνικό. Οι άνθρωποι πήγαιναν στη δουλειά τους, είχε πολλή κίνηση και πολλά από τα αυτοκίνητα με στην κίνηση είναι μεγάλα τζιπ ή πολυτελείς λιμουζίνες. Αναρωτιέται κανείς, πού βρίσκουν τα λεφτά τόσοι Ουκρανοί για να παίρνουν Λέξους και Mercedes. Και η απάντηση προέκυψε σε όλες τις συζητήσεις ε, που κάναμε. Διαφθορά, αχαλήνοτη. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, από ό,τι ακούσαμε, έχουν βουτήξει ε, λεφτά. Αλλά εκτός από την διαφθορά, αυτό που τους ανησυχεί είναι ο πόλεμος. Τους αποκαλούν ε, τρομοκράτες ή αυτούς που θέλουν να αποσχιστούν και λένε ότι κάθε μέρα καταπατούν την ε, κατάπαυση του πυρός και μας είπαν ότι αν η Ευρώπη δεν σταματήσει τη Ρωσία τότε ο στρατός του Πούτιν ε, θα φτάσει στα σύνορα της Ένωσης και θα τα διασχίσει. Μας είπαν επανειλημμένο ότι χρειάζονται επιγόντως όπλα, ότι ε, πολλές φορές ο, ο στρατός τους χρησιμοποιεί αρχαία όπλα. δεν έχουμε απαγορεύσει τη χορήγηση οπλισμού, αλλά δεν τους δίνουμε και οπλισμό. Έτσι λοιπόν ε, μάθαμε πολλά από αυτήν την επίσκεψη. Τουλάχιστον όμως εγώ έμαθα το εξής ένα. Εάν δώσουμε περισσότερα όπλα, στην ουσία θα παρατείνουμε τον πόλεμο και θα τον επεκτείνουμε κιόλας, Ενδεχομένω μέχρι τα σύνορά μας. 70 χρόνια μετά τη λήξη του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου αυτό είναι οπωσδήποτε κάτι που δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλες τις διπλωματικές δυνατότητες να σταματήσει η επιθετικότητα και να καταλάβει ο κύριος Πούτιν ότι αρκεί, όσο εδώ και μην παρέκει. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με το φίλο μου τον κύριο Γκάλαρ ότι φυσικά δεν πρέπει να έρθουν οι κυρώσεις και επίσης ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία της κυβέρνησης της Ουκρανίας να εισαγάγει μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Κύριε Πλένκοβιτς, ε, και εσείς ε, συμμετείχατε σε πολλές από τις συναντήσεις που κάναμε Πρόκειται για κοινή αποστολή μεταξύ τη Επιτροπή μα και τη Αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Ουκρανία. Οπότε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ω πρόεδρο τη Αντιπροσωπεία είναι πολύ καλό ότι από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλήσαμε με μία φωνή στα πλαίσια μία αντιπροσωπεία, ΣΕΝΤΕ, budget και εγώ μαζί από πλευρά αντιπροσωπεία. Νομίζω ότι είναι ένα σαφέ μήνυμα ότι μιλάμε με μια φωνή και ότι είναι συνέχιση της πρώτης μας συνάντησης στα πλαίσια της Επιτροπής Σύνδεσης. Ε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΕΝΤΕ, το πιο σημαντικό ήταν αυτά που ακούσαμε για την αποτελεσματικότητα του ρόλου της ειδική αποστολής του ΟΑΣΕ. Αυτά μας είπαν οι Ουκρανοί φίλοι, είπαν ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες βελτίωσης. Δεύτερον, υπάρχει σαφής επιθυμία της Ουκρανικής πλευράς να, να υπάρξει μια αποστολή της κοινή ε, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, όχι μόνο η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του μη στρατιωτικού τομέα. Για μένα αυτό ήταν σημείο κλειδί ότι θέλουν να υπάρξει αποστολή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και επίσης ενδιαφέρον είναι ότι η διαδικασία σταγματικής μεταρρύθμισης και αποκέντρωσης, ιδιαίτερα για τις ε, κατεχόμενες περιοχές του Ντομπάς, είναι προϋπόθεση. Όχι, αντίστροφα. Ότι για να γίνουν όλα αυτά πρέπει πρώτα να γίνουν έντιμες εκλογές. Μόνο μετά θα μπορέσει να γίνει αποκέντρωση. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, έμεσα να εγκρίνουμε τις παράνομες εκλογές στις περιοχές αυτές της ε, Δευτέρας Νοεμβρίου. Επίσης, είναι ενδιαφέρον το πώς οι διάφορες επιτροπές εκτιμούν διαφορετικά την κατάσταση πραγμάτων στη χώρα. Όταν πήγαμε στην ε, Ουκρανική Βουλή με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Άμυνας, εκεί είδαμε ότι προφανώς θεωρούνται ότι είναι σε κατάσταση πολέμου. Ήταν λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ακόμη και για μένα που πηγαίνω συχνά στην Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ για τη θαυμάσια συνεργασία όλης μας της αντιπροσωπείας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της αποστολής της ΕΝΤΕ και της αντιπροσωπείας. Συμφωνώ και συμμερίζομαι τις απόψεις σας ότι ήταν πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι και να διαβεβαιώσουμε τους Ουκρανούς συνομιλητές μας ότι το κοινοβούλιο μας τους υποστηρίζει σταθερά τη χώρα και το λαό. Είδαμε πολλά. Την ανθρωπιστική κατάσταση, τα κοινωνικά θέματα, συναντηθήκαμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις που φροντίζουν για τα εσωτερικά μετατοπισμένα άτομα και συνολικά θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτών των εσωτερικά μετατοπισμένων ατόμων είναι σχετικά εντάξει, δεν θα λέγα καλή βέβαια, επειδή υπάρχουν πολλές προσπάθειες από πλευράς των μη κυβερνητικών οργανώσεων και από την κοινωνία των πολιτών εντός της Ουκρανίας. Είναι πολύ παρούσα η κοινωνία των πολιτών σε τέτοια έκταση που τα καταφέρνουν όχι μόνο να βοηθήσουν αλλά να υποκαταστήσουν τις δημόσιες αρχές στην προσπάθεια αυτή. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ ευγνώμονες προς τις Ουκρανικές μη για τη δουλειά που κάνουν. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή μαζί τους και στο μέλλον. Για να δούμε πώς θα πάνε. Τώρα έχουμε τον ομιλητή για το επόμενο θέμα που είναι ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ που επρόκειτο να έρθει για το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο θα συζητήσουμε από κοινού με την ΑΦΕΤ για να ανταλλάξουμε απόψεις με τον κύριο Φρανκ Μπρένερ που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Eurocontrol. Είχαμε μια κοινή αποστολή, επισκεφθήκαμε το Eurocontrol πολύ πρόσφατα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπρένερ και τους συνεργάτες του Και τώρα να ακούσουμε τη δική του παρουσίαση στην υποεπιτροπή μας σε συνεργασία με την ΑΦΕΤ. Και ο δεύτερος συνομιλητής μας είναι ο κύριος Μπογκδάν Γκαϊεύσκι. ο οποίος είναι ένας ε, εξέχων ειδήμων της καναδικής κυβέρνησης υπεύθυνο για τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων. Το θέμα της συνάντησής μας είναι η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας σε περιοχές συγκρούσεων. και σε περιοχές που ελέγχονται από στρατιωτικές δυνάμεις. Και οι κίνδυνοι για την πολιτική αεροπορία που προκύπτουν, προκύπτουν από τις πτήσεις ε, μαχητικών. Να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΑΦΕΤ, τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Χαίρομαι που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε συγκεκριμένα ατυχήματα που προέκυψαν σε περιοχές όπου υπάρχουν κρίσεις και θέλουμε να δούμε με τι τρόπο μπορούν να συνεργάζονται περισσότερο οι οργανισμοί ελέγχου των πολιτικών ε, πτήσεων και των στρατιωτικών πτήσεων. Αυτό είναι θέμα και οικονομικής ε, σημασίας. Γιατί πολλές φορές ε, τα αεροπλάνα μας χρειάζεται να κάνουν zigzag πάνω από την Ευρώπη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνδυάσουμε καλύτερα τις εναέριες περιοχές για την πολιτική αεροπορία και για τη στρατιωτική αεροπορία. Ξέρουμε ότι αυξάνεται επίση γενικά η κυκλοφορία στους εθέρες, οπότε το θέμα αυτό έχει μεγάλη οικονομική σημασία. Και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να δώσω απευθεία το λόγο στον ε, Μπέρναρντ για να μας κάνει μια εισαγωγή. Σας ευχαριστώ για την ε, εισαγωγή που κάνετε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να σας μιλήσω για το τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα. Αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα χαρώ πολύ να μοιραστώ μαζί σας ε, την εμπειρία που έχω σε σχέση με την ε, κατάσταση προς την ε, ασφάλεια στον αέρα και την, τις τελευταίες εξελίξεις σε πόλεμες ζώνες, κυρίως σε σχέση με την ασφάλεια στα ανοιχτά της θάλασσας. Εκπροσωπώ το Eurocontrol, είναι μια διακυβερνητική οργάνωση με 41 κράτη-μέλη από την Ιρλανδία, μέχρι την Αρμενία. Α, και η Ουκρανία είναι μέλος μας, όπως βλέπετε. Ε, ε, επίσης, ε, το Εύρος πάει από την Πορτογαλία μέχρι την Εσθονία, στην κατεύθυνση νότος-βορράς. Είναι πανευρωπαϊκή λοιπόν η προσέγγιση και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την ασφάλεια για τη διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας διότι πετούν σε ολόκληρη την Ευρώπη τα αεροσκάφη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μιλάμε με μία ευρωπαϊκή φωνή και με τα, οι χώρες που δεν ανήκουν στην Ένωση ε, θα πρέπει να ε, παραμείνουν σε στενή συνεργασία μαζί μας. Σε αυτό αποσκοπούμε ούτως ώστε ε, να είμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή οργάνωση όπως και ο ΙΚΑΟ. Δεν είμαστε ευρωπαϊκός θεσμός, θεσμός Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως έχουμε μια υψηλό επίπεδο συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της οποίας συνεργαζόμαστε στενότατα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα όπως ο ΕΑΣΑ, παραδείγματος χάρη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας για την Αεροπορία, την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα εργασία. Εμείς είμαστε μια οργάνωση πολιτικής πολιτικο-στρατιωτική ε, με στόχο να συντονίζουμε τις διαφορετικές ανάγκες που έχει η πολιτική και η στρατιωτική αεροπορία σε έναν ενίο εναέριο χώρο. Ένα βασικός ρόλος ε, του Ευρωκοντρόλ είναι ο διαχειριστής του δικτύου. Διοριστήκαμε σε αυτό το ρόλο το 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκτοτε ε, χρησιμοποίησαμε την πρώτερη εμπειρία μας για την διαχείριση της ροής με ε, αναγνωρισμένη επιτυχία και δεν καλύπτουμε μόνο τον αέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών αλλά των 41 κρατών μελών του Eurocontrol ακόμη και πέραν αυτού διότι συνεργαζόμαστε και με χώρες όπως το Μαρόκο ή και άλλες γειτονικές μεσογειακές χώρες, ανταλλάσσουμε σχέδια πτήσεων, ενημερώσεις και στίγματα αεροσκαφών στον αέρα, ε, είτε πρόκειται για πολιτικά είτε για στρατιωτικά αεροσκάφη. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους ως προς επιδόσεις είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό τις καθυστερήσεις καθοδών ε, και μόνο λίγα δευτερόλεπτα, 30 συγκεκριμένα επιτρέπονται για κάθε πτήση. Ε, αν το πολλαπλασιάσετε αυτό με 30.000 πτήσεις την ημέρα ή 10 εκατομμύρια πτήσεις το χρόνο βλέπετε ότι είναι σχετικά δύσκολο να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος όμως προσπαθούμε να είμαστε τόσο ακριβείς και αυτά είναι τα καλά νέα. Ε, θα πρέπει να παραδεχτούμε επίσης ότι ο στόχος θα μπορούσαμε να τον υλοποιήσουμε στην Ευρώπη αν δεν υπήρχε στενή συνεργασία ανάμεσα στους χρήστες ε, του πολιτικού και στρατιωτικού ενερίου χώρου χρησιμοποιώντας αυτό που υπονομάζουμε ευέλικτη χρήση του εναερίου χώρου πρόκειται ε, για ένα ε, τομέα στον οποίο νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ανατεθεί η διαχείρισή του στο Ευρωκοντρόλ. Τα γεγονότα στην Κρυμαία και στην Ανατολική Ουκρανία έχουν οδηγήσει σε πολύ μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τα μοντέλα της ενέργειας κυκλοφορίας και υπάρχει συμφόρηση μεγάλη σε περιοχές όπως ε, ε, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία και βλέπετε πάνω πάνω στην εικόνα για το 2013 την Ουκρανία όπου βλέπετε πάνω από τον Εύξηνο Πόντο και την Ουκρανία πολύ ισχυρή ροή αεροσκαφών ξαφνικά στέγνωσαν αυτά και όλα έχουν μετατοπιστεί προς τον νότο όπως σας είπα στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στην ε, Τουρκία. Όχι περαιτέρω βεβαίως και θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα ότι έχουμε πολλούς περιορισμούς νοτιότερο. Συρία, Τουνισή, την Ισία, Λιβύη, οπότε ε, αυτή τη στιγμή δρομολογούμε όλα ανάμεσα σε αυτό το χώρο, ανάμεσα στη Μεσόγειο και τον Εύξηνο Πόντο και ε, γι' αυτό υπάρχει συμφόρηση στον εναέριο χώρο, δεν είναι καλό αυτό, όμως είναι απόρρια της τρέχουσας ε, πολιτικής κατάστασης. Αυτό αποκαλούμε διαχείριση του δικτύου σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και σε σχέση με τη διαθεσιμότητα τη της δυναμικότητας που έχουμε. Αυτός είναι ο ρόλος του διαχειριστή δικτύου. 24 ώρες το 24ωρο ε, προσαρμοζόμαστε στην, ε, στις εξελίξεις ε, ανάλογα με το αν ανοίγει η κλίνη κάποιος αέριος χώρος ή αεροδιάδρομος και αυτό θα πρέπει κυρίως μετά τις εξελίξεις του MH17 του αεροσκάφους των Malaysian Airlines διότι συνέβη αυτό το ατύχημα όταν άνοιξε ο ενέργειος χώρος και μπόρεσε το MH17 να πετάξει πάνω ε, από αυτό τον ενέριο χώρο. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες νόταμς, τις αγγελίες που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Έχουμε με μια παγκόσμια συμβέλεια σε βάση δεδομένων, συλλέγουμε τα δεδομένα και τα καθιστούμε διαθέσιμα σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλους τους αερομεταφορείς. Αυτές τις πληροφορίες ε, λοιπόν πρέπει να τις έχουμε στη διάθεσή μας. Όμως το θέμα είναι πώς ακριβώς ε, λαμβάνουμε την απόφαση. Πώς, πώς ακριβώς ε, ποια είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τι γίνεται λοιπόν από πλευράς του αερομεταφορέα. Κοιτάζουν τους αεροδιαδρόμους που είναι ανοιχτοί και βλέπουν ποια κριτήρια θα χρησιμοποιήσουν. Βλέπουν ε, ε, τον χρόνο, τις επτήσεις, ε, το καύσιμο, τις εκπομπές, τις αλλαγές στον καιρό, επίσης τον χρόνο άφηξης και πάνω από όλα, αλλά πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της ασφάλειας. Τώρα το θέμα είναι πώς μπορεί ένας ε, αερομεταφορές, ένα κράτος να αποτιμήσει την ασφάλεια γύρω από ένα αεροσκάφος στην Ευρώπη. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό, η υποχρέωση των κρατών μελών να ε, μεταβιβάζουν αυτές τις αποτιμήσεις της ασφάλειας κοιτάζουν ε, τον εναέριο χώρο και εξετάζουν την κατάσταση. Είναι ασφαλής μια πτήση σε εκείνη την περιοχή και το θέμα είναι αυτές οι πληροφορίες και οι εξολογήσεις να μην ε, παραμένουν μόνο στα χέρια τους, αλλά στο μέλλον σκοπούμε στο να υπάρχει διανομή αυτών των πληροφοριών. Μετά το MH17 συγκροτήθηκε μια task force και εντοπίσαμε ότι ε, κρίθηκε ασφαλής μια πτήση στην Ουκρανία του εκεί όπου έπεσε το MH17 ήταν πλημελής η αξιολόγηση, είναι προφανές, όμως δεν ήταν δυνατόν να το γνωρίζουμε αυτό διότι δεν κοινοποιήθηκε η αξιολόγηση σε σχέση με την ασφάλεια. Οπότε αυτή είναι και, και το βασικό τροτό σημείο του συστήματος μας ότι δεν κοινοποιούνται ανάμεσα στα κράτη-μέλη αυτές οι αξιολογήσεις για την ασφάλεια. Μετά το MH17 ε, στο Montreal ο ΕΚΑΟ ε, συγκρότησε μια task force και έκανε μία, πριν από λίγε εβδομάδες και μία διάσκεψη υψηλού επίπεδου για αυτό το ζήτημα και το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να καλύψουμε αυτή την έλλειψη του συστήματος και θα πρέπει να τροποποιήσουμε το σύστημα του στα κράτη-μέλη, ώστε να καθίστανται διαθέσιμε οι αξιολογήσει για την ασφάλεια. Έχουμε ένα παράδειγμα ε, στην ε, πράξη, έχει εφαρμοστεί αυτή η νέα αρχή, παραδείγματο χάρη το αεροδρόμιο του Τελαβίβ, όταν δέχτηκε πρόσφατα επίθεση με πυράβλους στα πλαίσια από την, που προέρχονταν από τη Γάζα, στα πλαίσια της ε, διαμάχης με τους ε, Παλαιστινίους. Σταμάτησε λοιπόν ένα αεροσκάφος, ε, την διέκοψε την πτήση και Υπήρξε και ενημέρωση από το Τελαβίδ προς τα Αμερικανικά αεροδρόμια για να ακυρωθούν οι πτήσεις και ακολουθήθηκε η συμβουλή και από την ευρωπαϊκή πλευρά από τον ΕΑΣΑ. Ε, κοινοποιήθηκε η πληροφορία για την ασφάλεια στο Τελαβίδ, έγινε αυτή η αξιολόγηση ε, και οι Αμερικανικές αρχές και ο ΕΑΣΑ ε, προγραμμάτισαν τις πτήσεις ε, τις, πάνω από το Τελαβίβ. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι το πλεονέκτημα όταν υπάρχει κοινοποίηση των πληροφοριών. Ο Ευρωκοντρόλ αυτή τη στιγμή θα τα κράτη-μέλη να γνωστοποιούν τις αποτιμήσεις κινδύνων σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά και σε όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου όπως πρόσφατα τους ενθάρρυνε ο ICAO. Εδώ βλέπετε την πληροφόρηση που έχουμε τώρα για το που υπάρχουν ε, περιοχές όπου έχει κλείσει ο αέρος χώρος, που υπάρχουν προειδοποιήσεις, τι πληροφόρηση υπάρχει και ποια είναι η βάση της αποτίμησης του κινδύνου. Με τι στοιχεία δηλαδή γίνεται. Μετά το MH17 και μετά τις συστάσεις του ICAO, το Eurocontrol, έχει φτιάξει ένα προστατευμένο τέτοιο σύστημα ούτως ώστε όλοι όσοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις να έχουν την αναγκαία πληροφόρηση. Οι χρήστες λοιπόν του εναέριου χώρου μπορούν να δουν τι κίνδυνοι υπάρχουν, πού είναι και πώς να αντιδράσουν στους κινδύνους. Αυτό το κάνουμε σταδιακά τώρα. Όλο και περισσότερα κράτη κοινοποιούν την πληροφόρηση που έχουν. Αυτό είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο να ληφθούν αποφάσεις, αλλά να έχουμε και τη βάση για την αποτίμηση του κινδύνου, αλλά να είναι συνεχώς ενημερωμένες αυτές οι ε, πληροφορήσεις. Πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς η εκτίμηση του κινδύνου. Ως ε, Eurocontrol συμβάλλουμε σε αυτή την ιδέα του ICAO παγκοσμίω. Δίνουμε στοιχεία με εστίαση κυρίως στην Ευρώπη γιατί έχουμε πρόσβαση στους οργανισμούς που έχουν αυτή την πληροφόρηση και αυτά τα συμμεριζόμεθα με όλα τα κράτη και με τον Οργανισμό ε, Πολιτικής Αεροπορίας στην Ευρώπη με προστατευμένη μορφή. Εδώ βλέπετε ένα, μορφή. Εδώ βλέπετε ένα slide όπου βλέπετε πού είναι οι περιορισμοί και πώς είναι η κατάσταση στη Συρία, τη Λιβύη κτλ. Δεν μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε παρά νότια τις πτήσεις και έχουμε περιορισμούς και στην Ουκρανία. Οπότε μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας πάνε Τώρα, οι πτήσεις επιτήρησης και οι πτήσεις στις ανοιχτές θάλασσες. Τους τελευταίους μήνες στην Ευρώπη έχουμε πολύ εντατικές επιχειρήσεις επιτήρησης στις ανοιχτές θάλασσες. Αυτό είναι ανησυχητικό για πολλά ευρωπαϊκά κράτη και συζητήθηκε φυσικά σε, διάφορες, ε, σε διάφορα φόρουμ και στο Κοινοβούλιο. Τα κράτη-μέλη του Eurocontrol, ιδίω στη Βαλτική, έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό εντός του Eurocontrol. για να υπάρχει ασφάλεια στις πτήσεις πάνω από τις ανοιχτές θάλασσες. Μας ζήτησαν τα κράτη-μέλη τον προηγούμενο Δεκέμβρη να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αλλά είχαμε παγώσει όλες τις επαφές μας με τη Ρωσία που δεν είναι μέλος του Eurocontrol μετά τα γεγονότα στην Κρυμαία. Μας ζητήθηκε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια τεχνική συζήτηση για να αυξηθεί η ασφάλεια στις ανοιχτές θάλασσες. Συμμορφωθήκαμε αυτό το αίτημα, καλέσαμε τον ΝΑΤΟ, τις Αμερικανικές ε, Ένοπλες Δυνάμεις, τα μέλη κράτη του Eurocontrol και τις οργανώσεις πολιτικής αεροπορίας του Eurocontrol να έρθουν στις Βρυξέλλες για να κάνουν μια τεχνική συζήτηση, για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Για πρώτη φορά η Ρωσία συμφώνησε να συμμετάσχει σε τέτοια συνάντηση και για να συζητήσουμε σε τεχνικό επίπεδο για την ασφάλεια στις ανοιχτές θάλασσες και τη βελτίωσή της. Είχαμε ευρεία συμμετοχή, έγινε αρχές του μήνα αυτή η συνάντηση, πολύ πρόσφατο λοιπόν, και θεωρώ ότι πολιτικά ως επέτυχε η χειρονομία που κάναμε προς τους Ρώσους γιατί όχι μόνο κάνουμε αυτή τη συνάντηση εργασίας, το workshop, αλλά και κατέληξε ότι οι διαδικασίες του ΙΚΑΟ που έχουμε για τις ανοιχτές θάλασσες από τη δεκαετία του 60, όπου τότε είχαμε πολύ λιγότερα ε, πολιτικά σκάφη, καταλήξαμε λοιπόν ότι δεν αρκούν αυτές οι, οι διατάξεις και κατέληξε η συνάντησή μας για μια σειρά συστάσεις για βελτίωση για τον ΙΚΑΟ. Και συμφωνήσαμε να γίνει μια δεύτερη τέτοια συνεδρίαση στο Παρίσι με τον ΙΚΑΟ, από τον ΙΚΑΟ, αυτό το μήνα. Και θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Παρά λοιπόν όλα τα προβλήματα, τις ανησυχίες για αυτές τις πτήσεις, καλά ναι έχουμε, υπάρχει μια τεχνική πλατφόρμα όπου μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας για αυτές τις πτήσεις πάνω από τις ανοιχτές θάλασσες. Είναι δύσκολο να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ακόμη επεισόδια και ατυχήματα. Πρέπει να αποφεύγονται πάση θυσία. Αλλά όταν συμβαίνουν, υποχρέωση της αεροπορικής κοινότητας είναι να τα αναλύει με κάθε λεπτομέρεια, να δει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, τι έπαιξε ρόλο και να δει πώς θα μπορούσε να αποφευχθεί στο μέλλον, ούτω ώστε η διαχείριση τη κυκλοφορίας να γίνει ασφαλέστερη. Πολλά μπορούμε να κάνουμε με την εξέλιξη των διαδικασιών ελέγχου της εναέρεσης κυκλοφορίας, πολιτικής και στρατιωτικής. Αυτά πρέπει να γίνονται μέσω ενημέρωσης όλων προς όλους. Αυτά τα έχει αναπτύξει και στο παρελθόν το Eurocontrol και τα έχει εφαρμόσει στην ομοθεσία της η Ένωση. Και δεσμεύουμε ενώπιον σας, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι είμαστε στη διάθεσή σας και γενικά του ευρωπαϊκού κοινού για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια γιατί έχει αποδώσει τα τελευταία 30 χρόνια. Υπάρχουμε εδώ και 50 χρόνια και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξουν σωστές διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορίας συμπεριλαμβανομένων και όλων των οργανώσεων που δεν συμμετέχουν στο Eurocontrol το 41 για το καλό των επιβατών. Ευχαριστούμε κύριε Μπρένα για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον δόκτωρα Μπόγκταν Γκαϊεύσκη και μετά κύριε Μπρόκ αν θέλετε να παρέμβετε μετά θα ανοίξουμε τη συζήτηση. My name is Bogdan Gajewski. My aviation background span... Ε, πάνω από 40 χρόνια έχω εμπειρία σε αυτό το τομέα και τα τελευταία 25 ε, χρόνια ε, είμαι ε, εκπρόσωπος του Καναδά με την ιδιότητα του μηχανικού. Ε, στο σχετικό φορέα της. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε ε, ε, τραγικές επιπτώσεις όλων των πολιτικών εξελίξεων. Ας πάρουμε την πρώτη περίπτωση Στις 22 Νοεμβρίου 2003 ένα κάργο Airbus ε, της, ε, του European Air Transport ε, χτυπήθηκε από πύραυλο της Ρωσίας. Οι δύο Βέλγοι και ένας Σκοτσέζος κατάφεραν παρόλα αυτά να προσγειώσουν το αεροσκάφος. Στη συνέχεια, 17 Ιουλίου 2014, το MH17 των Malaysian Airlines καταρρίφθηκε πάνω από την Ανατολική Ουκρανία και πέθαναν 298 άνθρωποι. Τρίτη περίπτωση, 10 Απριλίου 2010, ένα πολωνικό αεροσκάφος ε, ε, έπεσε στο Σμολένσκα και πέθαναν και οι 96 επιβάτες. Ε, φυσικά, λυπούμεθα για τις ζωές που χάθηκαν, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να επαναληφθούν στο μέλλον τέτοιες τραγωδίες και θα πρέπει να αντιλήσουμε τα διδάγματά μας από τις εκθέσεις σε σχέση με τα ατυχήματα. Για την τρίτη περίπτωση, TU-154M, δηλαδή το πολωνικό αεροσκάφος, προς το παρόν έχουμε μόνο μία διαθέσιμη έκθεση για αυτό το ατύχημα ε, και σχετίζεται με το ε, ατύχημα λοιπόν που έγινε στο Σμολένσκ στη Ρωσία όπου έπεσε αυτό το στρατιωτικό αεροσκάφος ε, και αυτό είναι το αντικείμενο της παρουσίασης μου. 10 Απριλίου 2010 το ένα πολωνικό TU-154M έπεσε κοντά στην πόλη του Σμολένσκ στη Ρωσία και πέθαναν και 96 επιβάτες μεταξύ των οποίων και πρόεδρος της Πολωνίας Ελέ Χατσίνσκι, η σύζυγός του Μαρία, ο πρώην πρόεδρος ε, Καζορόφσκι, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατού και άλλοι υψηλότατοι πολωνινοί αξιωματούχοι. 88 ήταν οι επιβάτες και το ε, ε, πλήρωμα ήταν 8 ε, άτομα. Από την Βαρσοβία ε, έφυγε ε, το αεροσκάφος και έπεσε στο Σμολένσκ. Αυτή ήταν η διαδρομή. Βλέπετε τώρα το, ε, στο Σμολένσκ την περιοχή του ατυχήματος. Η έρευνα που έγινε κατέληξε σε δύο επίσημες εκθέσεις. Η ρωσική έκθεση που φέρει τον τίτλο ΜΑΚ και η πολωνική έκθεση Μίλερ από το όνομα του συντάκτη κάθε φορά και έχουν ταξινομηθεί έχει ταξινομηθεί το ατύχημα ως ε, ελεγχόμενη πτήση ε, που προσκρούει στο έδαφος και από τις δύο εκθέσεις και συνήθως δηλαδή θεωρείται ότι πρόκειται για λάθος του πιλάτου. Βασική αρχή οποιασδήποτε έρευνα για ένα τέτοιο ατύχημα είναι ότι αν σημειωθούν διαφορές ανάμεσα στις δύο αντιπαραβαλλόμενες έκθεσεις θα πρέπει να, απορριφθεί, ε, να απορριφθούν και οι δύο εκθέσεις. Υπάρχουν βασικές ε, διαφορές ανάμεσα στις εκθέσεις και αυτό ε, μας οδηγεί στο να αμφιβάλλουμε για την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό με τον οποίο έγιναν αυτές οι έρευνες. Ε, ε, χρησιμοποιούνται μόνο βασικά στοιχεία και δεν μπορεί να επικυρωθεί η ποιότητα των εκθέσεων. Α πάρουμε τώρα τι πληροφορίε ε, για βασικού τομεί, όπω παραδείγματο χάρη η απογραφή που έγινε ε, επί τόπου, η διάταξη τη καμπίνα μέσα στο αεροσκάφο, η ώρα του ατυχήματο, το μαύρο κουτί και η έρευνα. Θα αρχίσουμε με το πρώτο. Η απογραφή που γίνεται επί τόπου έχει καταλητική σημασία για οποιαδήποτε τέτοια έρευνα και πρέπει να υπάρξει μια περίμετρος ασφαλείας, να υπάρξουν αλλαγές ε, επί τόπου. Αυτό δεν έγινε όμως σε συγκεκριμένη περίπτωση και ο ντόπιο πληθυσμός ε, μπόρεσε λοιπόν να έχει πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος αλλάζοντας τα τεκμήρια. Βλέπετε τρία τώρα παραδείγματα ε, αυτού που ισχυρίζομαι στις ε, φωτογραφίες αυτές. Βλέπετε επίσης στην αεροφωτογραφία ε, γίνεται ανταπαραβολή ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ε, χρονικές στιγμές και βλέπουμε ότι μετατοπίστηκαν τα συντρίμια του αεροσκάφους. Αυτό αναφέρεται στη δεύτερη εκθεσή. Πρόκειται κυρίως για το πίσω ωραίο πτέρωμα. Όπως έλεγα, μπόρεσε ο ντόπιο πληθυσμό να έχει πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματο. Ε, άλλαξαν τα τεκμήρια και βλέπουμε στι ε, δορυφορικέ αεροφωτογραφίε ότι άλλαξε και ο τόπο στον οποίο βρέθηκαν τα συντρίμια. Ε, δεν έχει καθοριστεί εξάλλου που ακριβώς προσέκρουσε στο έδαφος ε, το αεροσκάφος. Υπήρξαν TG-154 αεροσκάφη με κωδικούς αριθμούς 101 και 102 ε, το 101 ε, προς ε, στο έδαφος στο Σμόλενσκ και κάθε αεροσκάφος πρέπει να έχει ένα πιστοποιητικό ε, πτυτικής ικανότητα, ε, Ο κύριος Γκάλερ διακόπτη, συγγνώμη, θα ήθελα να υποβάλω ένα άμεσο ερώτημα στην ε, Πρόεδρο της Επιτροπής. Για ποιο λόγο ε, παρουσιάζεται αυτή η έκθεση, δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, δεν έχουμε συμφωνήσει για κάτι τέτοιο και πραγματικά ε, επί τώρα εξετάζουμε αυτό το σημείο. Στην ημερήσια διάταξη που αποφασίζουν οι συντονιστές δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Ξαφνικά ε, γιατί ε, προκύπτει αυτό το θέμα είναι μια εσωτερική πολωνική υπόθεση μου φαίνεται αυτό που βλέπουμε να εκτελήσεται μπροστά μας ε, και εγώ δεν προτίθεμαι να το επιτρέψω. Και εγώ θα μου έρθει μια ιδέα αύριο χωρίς να το συμφωνήσω με κανέναν να καλέσω όποιον μου έρθει. Ε, νομίζω ότι ε, υπάρχει παραβίαση της διαδικασίας. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι συντονιστές, εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων ε, τι πιστεύουν γι' αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Αυτή η η παρουσίαση είναι ε, μέσα στην ημερήσια διάταξη διότι εξετάζουμε το θέμα των απειλών κατά της πολιτικής αεροπορίας ε, που σε εμπόλεμες ζώνες και σε ε, περιοχές υποστρατιωτικό έλεγχο. Δεν είναι ένα πολωνικό που μια πολωνική υπόθεση όπως ισχυρίζεστε. Είναι τρεις οι περιπτώσεις ε, που αναφέρονται στην παρουσίαση και υπάρχουν στα έγγραφα της ε, συνεδρίασης. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γκαγεύσκη πως είναι ε, της σημασίας το να κάνουμε την αξιολόγηση και την αποτίμηση όλων των περιπτώσεων ε, έγινα παρουσίαση για το MH17 και ε, στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας προς ε, τους Ολλανδούς μέλη των οικογενειών των θυμάτων. Τώρα μιλάμε λοιπόν για την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία για διάφορα είδη πτήσεων. Δεν καταλαβαίνω, ε, ε, ο κύριος Μπρόκ θέλει να παρέμβει. Αγαπητοί κυρία συνάδελφοι, ο κύριος Μπρόκ, νομίζω ότι εδώ με αντιμετωπίζετε με λάθος τρόπο. Προσκλήθηκα για να συζητήσουμε συνολικά το θέμα της ασφάλειας πτήσεων σε περιοχές συγκρούσεων και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση γι' αυτό. Για αυτό το θέμα τώρα, να κάνουμε μια εσωτερική πολωνική συζήτηση που θέλει να αξιοποιήσει για προεκλογικό λόγο το κόμμα σας. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επανειλημμένα έχουμε πει ότι βεβαίως έχουμε κάθε συμπαράσταση μαζί σας και λυπούμεθα για τα θύματα του ατυχήματος στο Σμολένσκ, αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να δούμε τι οδήγησε σε αυτό το θέμα. Μπορεί να έχει κανείς πολύ διαφορετικές ε, απόψεις. Το θέμα είναι πώς θα πρέπει να διασφαλίσουμε οι περιοχές συγκρούσεων να μην αποτελούν κίνδυνο για την πολιτική αεροπορία. Και ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπρένα που υπέβαλε προτάσεις. Αλλά ως πρόεδρος της ΑΦΕΤ δεν είμαι διατεθειμένος να συμμετάσχω σε μια εσωτερική πολωνική αντιπαράθεση. Εντάξει, τώρα μπορεί να έρθει από το κόμμα σας να πάρουν το λόγο όλοι, αλλά σας παρακαλώ να μην κάνετε κατάχρηση των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό παρακαλώ τον συνάδελφο Μπαγεύσκη να καταλήξει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη γενικότερη συζήτηση. Παρακαλώ. Μου επιτρέπετε θα ήθελα να απαντήσω στις ε, κατηγορίες ε, του Πρόεδρου της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Όπως φαίνεται, η επίθεση της Ρώσικης Ομοσπονδίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναθεώρηση πολλών αποφάσεων και συμπερασμάτων που αφορούν για παράδειγμα τόσο συνέψαν στη Γεωργία θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αναθεώρηση της έκθεσης του πρέσβη ως προς το ποιος ήταν ο επιθέμενος και ποιο το θύμα. Κοιτώντας ε, τις διάφορες αυτές ε, περιπτώσεις ε, και κοιτώντας τα όσα βλέπουμε τώρα, την κατάληψη της Αυχαζίας και της Οσετίας, ε, ταυτόχρονα θεωρούμε ότι πρέπει να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε τι έχει γίνει με άλλα ε, συμβάντα όπως ε, το ατύχημα του Σμολένσκ. Δεν είμαι υποψηφίος σε κάτι κύριε. Δεν, είμαι, δεν είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής της Πολωνίας. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η παρουσίαση αυτή. Αν, αν εσείς αξιότιμα μέλη θεωρείτε ότι πρέπει να διακόψουμε τώρα αυτή την παρουσίαση μπορούμε να τη διακόψουμε, αλλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα είχε οποιοδήποτε ε, καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ως πρόεδρος της ΑΦΕΤ παρακαλώ τον κύριο Καγεύσκη να τελειώσει την παρουσίασή του στα επόμενα 2-3 λεπτά. Παρακαλώ, τελειώνετε. Σε 2-3 λεπτά. Ε, εντάξει, θα προσπαθήσω να καταλήξω όσο ταχύτερα γίνεται. Να πάω κατευθείαν στα συμπεράσματα. Να δείτε πώς είναι ένα συνήθις ε, πύργος ελέγχου, όπως το βλέπουν οι ταξιδιώτες, και πώς είναι ο πύργος ελέγχου του στρατιωτικού αεροδρομίου του Σμαλένσκ. Πορίσματα. Και οι δύο εκθέσεις δεν τηρούν τις προδιαγραφές σε βάθος εξέτασης και υπάρχουν σοβαρές διαφορές στις εκθέσεις οι οποίες θέτουν να αμφιβόλο την ευσυνειδησία και τη σοβαρότητα των ερευνητών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκαϊεύσκη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχω σημειώσει τα αιτήματα. Ε, κύριε Γκάλαρ, θέλετε να λάβετε το λόγο ως συντονιστής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπρένερ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Ε, σας έχω δει και ε, στο αεροδρόμιο προηγουμένως. Για μένα είναι σημαντικό ότι ο οργανισμός ε, Eurocontrol πρέπει να είναι το κέντρο και η σαφής απόδειξη ότι μπορούμε να συνεργαστούμε διαμεθοριακά για να καταλήξουμε στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Αυτό είναι πολιτικά το αποφασιστικό, αξιοποιώντας τις εμπειρίες των διαφόρων κρατών μελών που ήδη συνδυάζουν την πολιτική και στρατιωτική εναέρια κυκλοφορία για να αυξηθεί η ασφάλεια των πτήσεων να μην είναι δηλαδή δύο διαφορετικοί κόσμοι που δεν επικοινωνούν ενώ λειτουργούν ένα δίπλα στον άλλον γιατί ο ενέργειος χώρος είναι ένας πρέπει λοιπόν να συνεργάζονται γιατί έτσι κερδίζουμε και χρόνο και χρήμα γιατί μπορούν ορισμένες πτήσεις λοιπόν να γίνουν χωρίς παρεκκλήσεις χωρίς τεφλασμένες γιατί κάποια τμήματα του αέριου χώρου είναι κλειστά και σε τελευταία ανάλυση το βασικό είναι σε τι βαθμό υπάρχει πολιτική βούληση από πλευρά των κρατών μελών, γιατί τα κράτη-μέλη πρέπει να συμφωνήσουν σε τελευταία ανάλυση για να υπάρξει πραγματικά ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Και θεωρώ ότι ο οργανισμός Eurocontrol είναι σημαντικός εταίρος μας, ήδη εργάζεται σε αυτό το τομέα. Το πολιτικό θέμα ή το θέμα προς εσάς θα ήταν ποια είναι η το θεμα προς θα ηταν ποια ειναι η συμβουλη σας, ποια είναι η σύστασή σας. Προς τις κυβερνήσεις που συναποφασίζουν και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το επιτύχουν αυτό. Εάν εσείς θέλατε να επιτύχετε αυτούς τους ανοιχτούς ουρανούς, ποια θα ήταν η πρότασή σας γιατί είστε εμπειρογνώμων για να την ακολουθήσουμε εμείς ως πολιτική. Πρόεδρος, ο κύριος Κάννα. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον ε, ε, αξιότιμο προσκεκλημένο για την παρουσίαση. Είναι πολύ ενδιαφέρον το μέσα αυτός. Διαρκώς ε, αυξάνεται η ενέργεια κυκλοφορία και οι στρατιωτικές δράσεις. Συνεπώς, το να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης είναι κρίσιμη σημασία. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Δεν ξέρω αν μια χώρα είναι καλό πράγμα, αλλά υπάρχει ανάγκη να γίνεται παγκοσμίω αυτό, έτσι δεν είναι. Και δεύτερον, είχαμε το ατύχημα των μαλαισιανών αερογραμμών. Πώ συνέβη αυτό, πώ γίνεται να μην γνωρίζουμε ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο και τι διδάγματα αποκομίσαμε από αυτό. Ευχαριστούμε, ο κ. Στάνοκ. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω δεδομένων των όσων συνέβησαν με τις μαλαισιανές ε, αερογραμμές ε, που έπεσαν ξαφνικά από τον ουρανό πάνω στην Ανατολική Ουκρανία και μετά από τις εσχρές προσπάθειες της προπαγάνδας στη Μόσχα να παραποιήσουν τα όσα συνέβησαν εκτίμησε ιδιαίτερα την παρουσίαση του κ. Γκαγιευσκή που μας δίνει μια γεύση του τι μπορεί να συνέβη και στο Σμολένσκα όπου πήραξαν κάποιοι τα τεκμήρια. Δεν είχα ξαναδεί τις ε, δορυφορικές φωτογραφίες και αυτό μας δίνει μια εικόνα του τι είναι ικανή να κάνει η Ρωσία για να καλύψει εγκληματικές πράξεις ή ε, την ανικανότητά της και τα δύο. Ε, το θέμα είναι ότι όλα τα τεκμήρια που υπήρξαν δείχνουν ότι στην Ουκρανία. Χρησιμοποιήθηκε ένα πυροβολικό σύστημα ρωσικό ε, τύπου μπουκ. Η Eurocontrol ενημερώνεται τακτικά από τις υπηρεσίες πληροφοριών, από τις συμμάχους των ΝΑΤΟ και από λοιπούς ε, για το κατά πόσο τέτοια συστήματα πέφτουν στα χέρια τρομοκρατικών ομάδων, γιατί σαφώς μόνο λίγες χώρες ε, περιλαμβάνουν τέτοια πυροβολικά συστήματα γης αέρος που μπορούν να φτάσουν σε ψώμετρο. Ελάχιστε χώρε κάποια μέλη του ΝΕΤ, ΝΑΤΟ, ίσω η Κίνα, η Ιαπωνία, είναι εξαιρετικά ακριβά μηχανήματα και εξαιρετικά επικίνδυνα και αν πέσουν σε λάθος χέρια. Και αυτό που με ανησυχεί, κάποια στιγμή, ξέρετε, προγραμματίζω να πάω στο Ερμπίλ, στο Κορδιστάν και είδα σε ένα χάρτη ότι ο αεροδιαδρόμος περνάει ακριβώς πάνω από ε, τα εδάφη που έχει καταλάβει το ISIS ε, στο Ιράκ. Και ε, τα μέλη έχουν ε, κλέψει πολύ εξοπλισμό. Έχουν κλέψει τέτοιο εξοπλισμό. Υπάρχει κίνδυνο να πετάει κανεί ε, πάνω από το Βόρειο Ιράκ και τη Βόρεια Ευχαριστούμε, Πάνκρα Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να πω ότι αισθάνομαι προσβεβλημένο που δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο κ. Γκαϊεύσκη με την παρουσίασή του. Ε, πιστεύω ότι εδώ αγγίζουμε το τη λογοκρισία. Φυσικά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε οριστικά τις αιτίε ε, της καταστροφής στο Σμόλενσκ, ε, δεν διευκρινίστηκαν. Ξέρουμε ότι έκλεισε το αεροδρόμιο. Ε, είναι και αυτό μια πτυχή που ανέφερε ο κύριος Μπρένερ. Αλλά αυτό που θέλω να πω κατά τη συζήτηση ακούσαμε ε, τους συναδέλφους να καταφέρονται επικριτικά κατά τη προπαγάνδα του Πούτιν. Αλλά όταν μιλάμε για το Σμόλενσκ ε, και, μετά λέμε ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ. Ε, δηλαδή τι κάνουμε. Δεν θέλουμε να συζητήσουμε κάτι το οποίο εμεί επικρίναμε στην προηγούμενη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να αναφερθώ ε, στα σημεία που είχαμε στην ημερήσια διαταξή σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την ασφαλεία των πτήσεων πάνω από εμπόλεμες περιοχές και οι περιοχές που ελέγχονται από στρατιωτικές δυνάμεις. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για την κατάρρευση της φύσης των Μαλισιανών αερογραμμών της φύσης 17. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι καταρρίφθηκε το αεροπλάνο αυτό. Έχουμε συζητήσει ήδη αυτό το ζήτημα και παρόμοια ζητήματα και βάσει των πληροφοριών που έχουμε λάβει από την ηγεσία της Eurocontrol ε, μας ανησυχούν διότι σε θέματα ασφάλειας στον αέρα, ασφάλειας για τα πολιτικά αεροσκάφη όπως φαίνεται οι πληροφορίες αυτές ε, ε, προέρχονταν ε, παλιά ε, από επιμέρους κράτη και παρέ, συγγνώμη, παρέμεναν σε επιμέρους κράτη και αυτό συνέβη και για αυτό το συγκεκριμένο αεροσκάφος οι Ουκρανικές αρχές δεν ενημέρωσαν ότι υπήρχαν τέτοιοι πύραυλοι στην περιοχή και τέτοια δυνατότητα κατάρριψαν ένας αεροσκάφους. Αναρωτιέμαι λοιπόν ε, στην Eurocontrol ε, χρησιμοποιείτε ακόμη τέτοιες πληροφορίες από επιμέρους χώρες και βασίζεται σε αυτές ή πραγματοποιείτε κάποια δική σας ανάλυση ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες ε, για να κάνετε μια τέτοια ανάλυση και αξιολόγηση. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερον, από τις πληροφορίες που ακούσαμε, κανείς δεν αναφέρθηκε στην ασφάλεια των αεροδρομίων και των αεροσκαφών όσον αφορά τα drones, τα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη, τα μη επανδρομένα. Μάθαμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει υπάρχει κίνδυνο ε, πρόσκληση ε, τηλεκατευθυνόμενων ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών σε αεροδρόμια, όπω έγινε πέρσι στο Heathrow. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για drones αστικής χρήση, αλλά και για στρατιωτικά. Θα ήθελα λοιπόν να μα δώσετε κάποιε παραπάνω πληροφορίε γι' αυτό είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ρυθμίζουμε εδώ στην Ευρώπη. Και αφού δεν το ρυθμίζουμε, ίσω να επέκειται ε, σύντομα κάποια σύγκρουση με εκατοντάδες ε, θύματα. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Μπροκ. Μέση Μπροκ. Ευχαριστώ για αυτά περί λογοκρισία. Νομίζω ότι ο κύριος Γαλεύσκη Ε, είχε αρκετό χρόνο να μιλήσει παρά το ότι δεν υπήρχε θέμα στην ημερήσια διάταξη. Εμείς θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά τους ελέγχους αέρες κυκλοφορίας για να μην ε, προκύπτουν γεγονότα όπως η κατάρριψη του MH17. Αυτός νόμιζα πως ήταν ε, ο τίτλος του θέματος της ημερήσιας διάταξης και καλέσαμε ένα οργανισμό που συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Ε, υπάρχουν προβλήματα που ε, που, που ε, διαφεύγουν από τις ε, ε, αρμοδιότητες του Eurocontrol. Για παράδειγμα, η περιοχή του Αρμπίλ. Πήγα από τη Βαγδάτη πίσω στην Ευρώπη μέσω του Αρμπίλ. Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Όταν βλέπει κανείς τι γίνεται, αυτά φοβίζουν. Τις τελευταίες εβδομάδες οι αυστριακέ αυστριακές αερογραμμές σταμάτησαν τις πτήσεις τους προς, προς το Αρμπίλ. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα των τηλεκατευθυνωμένων αεροσκαφών, των drone. Όποιος έχει ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην Ουκρανία, να ανέβει μέχρι κάποιο, κάποιο υψόμετρο και πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για να ε, ελέγχουμε ε, αν είναι κοντά σε ένα αεροσκάφο, σε ένα τέτοιο ντρόουν για να μπορούμε να ενημερώσουμε τα αεροσκάφη. Επίσης, υπάρχουν ε, επίσης φορητές, φορητά όπλα κατάρτισης αεροσκαφών. είναι δυνατόν αν πετάμε πολύ ψηλά να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο. Γιατί αυτά τα ε, αυτά τα όπλα μπορούν να εκτοξεύσουν πυράβλους μέχρι 6-7 μέτρα. Πρέπει λοιπόν να πετάμε πάρα πολύ ψηλά. Σε ορισμένε περιπτώσει όμω προσέγγιση ε, μπορούν τέτοια φορητά όπλα να χτυπήσουν αεροσκάφη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είναι δύσκολο το Ισλαμικό κράτος να πάρει drone, να αποκτήσει drone ή άλλα τέτοια φορητά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αν ασχοληθούμε με το θέμα της Ουκρανίας και με την Μέση Ανατολή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο τείχος που θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο ακριβή την ε, ένα κυκλοφορία, τις πτήσεις δηλαδή, και ίσως για ορισμένα πράγματα θα πρέπει να πετάμε πάνω από τους πόλους για να πάμε από τη μια μεριά του κόσμου στην άλλη. Εντάξει, είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Αλλά πέστε μου, είναι όντως υπερβολικό ή είναι ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Αν δεν θέλουμε οι επιβάτες μας των πολιτικών πτήσεων να κινδυνεύουν πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τανέτσκι. Σα ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς τον κύριο Γκαγιέσκη. Ως μέλος Επιτροπής, Υποεπιτροπής ε, ΣΕΝΤΕ θα ήθελα να ρωτήσω ποιες διατάξεις ε, των κανονισμών ΙΚΑΟ παραβιάστηκαν από τους δρόσους τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται ότι αυτές οι παραβιάσεις των διεθνών διατάξεων που έχουν επικυρωθεί από όλους μπορούν να επαναληφθούν και σε ποιο βαθμό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω το ερώτημά μου και στους, ε, στα δύο μέλη του πάνελ μας. Κύριε Μπρένερ, μας μιλήσατε για στρατιωτικές πτήσεις στα νυχτά της θάλασσας. Ε, και είναι πραγματικό πρόβλημα όταν πρόκειται για εμπόλεμες ζώνες. Ε, συχνά επίσης παραβιάζεται ενέριος χώρος πολλών κρατών, όχι μόνο κρατών μελών. Υπήρξαν πολλά τέτοια περιστατικά όπου παραβιάζουν συχνά τα στρατιωτικά αεροσκάφη τον ε, αέριο χώρο και ε, συζητούν απειλή για την ε, πολιτική αεροπορία. Σε μία επιτροπή της ΣΕΔΕ με μέλη της Λιθουανικής, Λετωνικής Αεροπορίας μας είπαν ότι καθημερινά έχουν τέτοιες παραβιάσεις. Επίσης ε, ε, ενημερωθήκαμε ε, ότι ακόμη και στην Πορτογαλία έχουμε τέτοια περιστατικά. Η κυρία Γκόμες μας ενημέρωσε μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα. Μπορείτε να μας πείτε σε επίπεδο Ευρωκοντρόλ κύριε Γαγεύση, ή ε, σε πλαίσιο κάποιων άλλων φορέων, ποια μέτρα θα μπορούσαν να αναλυφθούν για να γίνει μια αξιολόγηση και πρόληψη στην καλύτερη περίπτωση αυτών των περιπτώσεων. Ο κύριος Μπρόκ, νομίζω. Ναι, είναι πολύ σημαντική η ερώτηση. Το ότι ρωσικά μαχητικά έχουν κλειστά τα μηχανήματα αναγνώρισής τους. Αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος. Μπορούμε να τα δούμε στο ραντάρ. Μπορούμε να στείλουμε αεροσκάφη να τα, γνω... να τα γνωρίσουμε. Ή... Επειδή είναι τόσο ε, ταχαία αυτά τα αεροσκάφη, είναι κίνδυνος. Αυτό είναι απαράδεκτο από πλευρά της Ρωσίας. Είναι απαράδεκτο να έχουν κλειστά τα transponder του τα αεροπλάνα αυτά. Και άλλη συμπληρωματική ερώτηση. Ευτυχώ που συμμετέχει σε αυτή την τεχνική επιτροπή η Ρωσία. Θα υπάρξουν κανόνε ω κατάληξη. Τι πρακτικέ συνέπειε θα έχει η συνεδρίασή σα. Καλό είναι που συνεδριάσατε, ότι θα ξαναβρεθείτε σε μερικέ εβδομάδε, αλλά σύντομα θα έχουμε πρακτικέ επιπτώσει. Ούτω ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος. Thank you. There are no other, other requests. Ευχαριστούμε. Δεν ζητάει κανεί άλλο το λόγο, οπότε να ζητήσω από τον κύριο Μπρονόρ και μετά τον κύριο Γκριεύσκη να απαντήσουν. Α, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, έχω μια δεύτερη ερώτηση και είναι σημαντική. Σχετίζεται με αυτά που είπε ο κύριος Μπρόκ. Από την εμπειρία σας, θα καταφέρει η Eurocontrol να διατηρήσει αξιόπιστες ε, πληροφορίες ε, και πώς, ώστε να στηρίζει τις αποφάσεις της. Θα υπάρξει και ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων αν χρειαστεί, αλλά τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Μπράναρ και μετά τον κύριο Γκέγευσκη να απαντήσουν. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για το ενδιαφέρον σας για το ζήτημα. Θα προσπαθήσω πρώτα να απαντήσω το ερώτημα του κυρίου Γκάλα για το ποια θα είναι τα άμεσα μελλοντικά βήματα και πώς θα εξελιχθούν τα ευρωπαϊκά ζητήματα το 2011, όπως εξήγησα, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη ορίσε την Eurocontrol ως διαχειριστή δικτύου. Αυτή η, απόφαση ε, θεωρήθηκε ε, τεράστια επιτυχία αν ρωτήσετε τα αεροδρόμια και όλους τους διάφορους φόρους, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη πολλές προκλήσεις. Ωστόσο υπάρχει και ένα σημαντικό μια σημαντική πολιτική συνιστόσα. Πολλέ διαφορετικέ απόψει υπάρχουν για το πώ θα πρέπει να εξελιχθεί η διαχείριση του δικτύου. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να είναι καθαρά εμπορική δραστηριότητα στην αγορά και άλλε απόψει λένε ότι πρέπει να είναι μια δημόσια υπηρεσία ε, δομημένη για να χρησιμοποιηθεί ω τέτοια στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια του 2015 αναμένουμε να ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος για τον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό ΣΕΣ δύο ΣΥΝ μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και μετά θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το ΣΕΣ 2+. Εμείς προτείνουμε να διατηρηθεί ο διαχειριστής δικτύου ως αξιόπιστο ουδέτερη δομή. Αντιλαμβανόμαστε το επιχείρημα ότι δεν πρέπει να αποτελέσει μονοπόλιο για πάντα και ότι πρέπει να εισαχθούν και εμπορικά στοιχεία. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι να κάνουμε μια πρόταση στο Συμβούλιο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς εσάς το Κοινοβούλιο να σας προτείνουμε λοιπόν κάποιο είδους ίσως μεικτής δομής, δηλαδή να λέμε ότι υπάρχει μια στρώση δημόσιας ε, υπηρεσίας ε, εκ μέρους των κρατών μελών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, κομισιόν αλλά να υπάρξει και μια σειρά εμπορικών τεχνικών υπηρεσιών ώστε να ε, υποστηριχθεί και αυτή η πτυχή ε, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Αυτά πρόκειται να γίνουν. Θεωρούμε ότι η διαχείριση του δικτύου βρίσκεται ακόμα σε αρχική φάση. Πολλές προκλήσεις δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί. Αλλά, ξέρετε, σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου μαζιλεύουν. Γιατί δεν έχουν κάτι αντίστοιχο κάποιον οργανισμό που να συντονίζει τις ε, δραστηριότητες. Ίσως λοιπόν να μην τα έχουμε επιτύχει όλα, να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε γύρω μας, αλλά βρισκόμαστε σε καλή θέση. Όσον αφορά τις διαδικασίες του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, πιστεύω είναι σημαντικό να υπάρξει νομοθεσία που θα καταστήσει υποχρεωτικέ και για τα 28 κράτη-μέλη της διαδικασίας του Ενίου ευρωπαϊκού ουρανού. Και είναι σημαντικό και οι χώρες πέραν τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθούν τα ωφέλη αυτών των διαδικασιών και να τις ε, ε, αποδεχθούν είτε μέσω διμερών ε, συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εθελοντικά. Αλλά για εμά την Eurocontrol μια καταγερματισμένη προσέγγιση θα ήταν καταστρεπτική, διότι όσοι βρισκόνται εκτό Ευρώπη θα έκαναν κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι κάνουμε εμεί. Για παράδειγμα, η Τουρκία πέρυσι υιοθέτησε την ευέλικτη χρήση του εναέριου χώρου που σας έδειξα εθελοντικά, διότι αντιλήφθηκαν τα ωφέλη της. Και όταν μας ρώτησαν γιατί το κάναμε αυτό ε, διότι έχει νόημα, ενισχύει την Ευρώπη και η Τουρκία μέσω της Eurocontrol συμμετείχε στην ανάπτυξη αυτών των διαδικασιών λοιπόν για ποιο λόγο να μην τις υιοθετήσουμε αυτοί είναι λοιπόν μηχανισμοί τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιούμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον στο πλαίσιο μια δομημένη προσέγγιση, μέσω της οποία μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και την επιρροή τη Ευρώπη μέσω αυτών των κανόνων. Όχι λοιπόν δηλαδή να εστιαζόμαστε μόνο σε 28 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα. Η Γεωργία αναφέρθηκε. Είναι πολιτικά πολύ σημαντικό να είναι μέλο τη Eurocontrol η Γεωργία, να είναι στενά συνδεδεμένη με το σύστημα τη Eurocontrol και μέλο ουσιαστικά τη οικογένειά μα. Ένα παράδειγμα απλά είναι η Γεωργία. Πιστεύω λοιπόν ότι η με περαιτέρω Διαδικασίε έλεγχου και περαιτέρω ιδέε για να ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κατακαιρματισμού είναι δυνατή. Ε, πολλές τεχνικές λύσεις υπάρχουν που μπορούν να μετατραπούν σε νομοθεσία στο εγγύς μέλλον, αλλά να μην ξεχνάμε τις χώρες πέραν των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτές πρέπει να δεχθούν ε, αυτές τις διαδικασίες. Έχουμε δύο θέματα με τις μαλαισιανές γραμμές, ε, την κατάρρευση του αεροσκάφους για την οποία μιλήσαμε, αλλά έχουμε και το εξαφανισμένο αεροπλάνο, το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί. Ασχοληθήκαμε και με αυτό και είπαμε στο μέλλον δεν μπορούμε να δεχθούμε να χάνεται ένα αεροσκάφος και να έχει περάσει ένα έτος και να μην υπάρχει ίχνος. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις δυνατότητες ειχνηλάτησης των αεροσκαφών ε, τις δυνατότητες κοινή χρήση των δορυφορικών ε, πληροφοριών και των πληροφοριών ραντάρ που αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει ώστε να γνωρίζουμε μόνιμα που βρίσκεται κάθε αεροσκάφος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλύτερη κάλυψη ραντάρ στην Ευρώπη από τις άλλα μέρη του κόσμου αλλά υπάρχουν μέρη όπου η παρακολούθηση μέσω ραντάρ και δορυφόρων δεν είναι τέλεια. Είναι ζητήματα λοιπόν ε, αυτά που αφορούν τη... Ναι, το θέμα του να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο δεδομένων όπου να έχουν προσδοσία όλα τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουμε τη βιότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε τις πληροφορίες ε, ραντάρ των διαφορών χωρών ώστε να έχουμε μια γενική εικόνα όπου δεν υπάρχουν κενό. Ε, όπως ε, υπόθηκε με μια σύσταση του ΙΚΑΟ μέσω μια τέτοια συγκέντρωση πληροφοριών θα βελτιώσουμε την ποιότητα και θα καλύψουμε τα κενά. Είναι κάτι το οποίο ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων και τις παραβιάσεις, η κατάσταση έχει αλλάξει. Πριν από μερικά χρόνια η απειλή που υπήρχε ήταν κατά βάση ε, πύραυλοι που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τρομοκρατικές επιθέσεις. Και όπω είπε ε, ο κ. Μπρόκ, όμω εκείνοι οι πυραυλοί μπορούσαν να φτάσουν μόνο μέχρι συγκεκριμένο υψόμετρο και υπήρχε συγκεκριμένη επιτήρηση ώστε ε, πύραυλοι που κουβαλούσαν κάποιο στον νόμο του να μην μπορούν να αποτελέσουν απειλή για αεροδρόμια. Αλλά αυτό που συνέβη με τι μαλλισιανέ αερογραμμέ ήταν ένα θέμα ε, πληροφοριών. Πληροφορίε που κάποιοι γνώριζαν περισσότερο από άλλου. Η Ουκρανία δεν γνώριζε τα όπλα αυτά και έκρινε λάθο. Ε, και έτσι κράτησε ανοιχτό τον αέριο τη χώρο. Το σύστημα που σα έδειξα εγώ είναι μια προσπάθεια πρώτα απ' όλα να λαμβάνουμε όλες τις εθνικές πληροφορίες με την αξιολόγηση κινδύνων Πράγματα που δεν μοιραζόμασταν μέχρι σήμερα και αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Δεύτερον, θα προσθέσουμε μια δεύτερη πηγή πληροφοριών. Κάτι πολύ πιο δύσκολο φυσικά, επειδή όλε αυτέ οι πληροφορίε. Ε, δεν ε, είναι κοινέ για όλου απαραίτητα. Αλλά κάποιε πληροφορίε ήδη κυκλοφορούν σε εθνικό επίπεδο, τι οποίε ενσωματώνουμε αυτή τη στιγμή στο σύστημα. Μετά από τη ατύχημα των Μαλαισιανών, την κατάρρευση των Μαλαισιανών ε, αερογραμμών, όλο και περισσότερα κράτη είναι όλο και πιο διατεθειμένοι να μοιραστούν ε, κάποιε πληροφορίε σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί πλήρω όχι στην έκταση που θα θέλαμε, αλλά είναι σε εξέλιξη και σίγουρα το Κοινοβούλιο μπορεί να ενισχύσει και μέσω νομοθεσίας ε, ε, ώστε να ζητήσει, να αναγκάσει τα κράτη-μέλη να καταστήσουν διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες που ο ΙΚΑΟ είναι ο μόνος που μπορεί να ζητήσει αυτή τη στιγμή και μόνο εθελοντικά. Πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Η ΆΣΑ λειτουργεί και προς την ίδια κατεύθυνση ε, Παραλαβει ε, σύλλογη αυτών των πληροφοριών και αξιολόγηση με ένα ε, επιχειρησιακό τμήμα το οποίο συγκεντρώνει τι πληροφορίε και τι καθιστά διαθέσιμε. Υπάρχει λοιπόν κάποια συνεργασία. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν όμω ακόμη περισσότερα, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ουσιαστικά, όπω βλέπουμε στου χάρτε, ο ενέργειο χώρο που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή σε σχέση με το παρελθόν είναι πολύ μικρότερο. Και η αύξηση του αριθμού των πτήσεων δεν βοηθά ειδικότερα όταν πρέπει να δρομολογήσουμε πτήσει μέσω διάβλων πολυσθενών. Αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, χρησιμοποιώντα από κοινού πληροφορίε με τα κράτη-μέλη. Για το ζήτημα των μη επανδρομένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών βρισκόμαστε στην αρχική φάση μιας εντελώ ε, εξέλιξη. Οι εμπορικέ προβλέψει ε, δείχνουν ότι η αγορά αυτή θα επεκτείνει θα σημειώσει τεράστια ανάπτυξη στο μέλλον και για στρατιωτική και για πολιτική χρήση. Βρισκόμαστε λοιπόν στα πρώτα βήματα αυτής της τεχνολογίας και μελετάμε τώρα πώς ε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία. Έχουμε ε, τη στρατιωτική, τέτοια τεχνολογία και την ε, πολιτική, πρέπει να δούμε σε τι ψώμετρα θα χρησιμοποιούνται. Έχει ζητηθεί από την Eurocontrol πέρυσι στην Κομισιόν ε, ένας οδικός χάρτης για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ο οδικός χάρτης αυτός χρησιμοποιήθηκε στην πρόσφατη στη Ρήγα από την Επιτροπή για περαιτέρω συγκεκριμένα βήματα. Οι εργασίες λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά αυτή τη στιγμή οι τεχνολογικές λύσεις κατά κάποιο τρόπο εξελίσσονται πιο γρήγορα από ότι το νομοθετικό κομμάτι και το κανονιστικό κομμάτι. Εκεί βρισκόμαστε. Σε τελική ανάλυση αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εντείνουμε τις δραστηριότητε μας, τις εργασίες μας, ώστε να μπορέσουμε να παραμείνουμε ε, σε παρομοιβηματισμό με την εξέλιξη αυτής της αγοράς. Ε, αν πρόκειται για ε, μη στρατητική χρήση, μόνο εδώ στην Ευρώπη μπορούμε εύκολα να ασχοληθούμε με αυτό. Ε, έχουμε αρκετέ προφορίε για να αποφύγουμε, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να αποφύγουμε επικίνδυνα περιστατικά όπω το χήθρο όπω αναφέρθηκε. Για τι περιπτώσει τρελατική χρήση ε, το ζήτημα είναι εντελώ διαφορετικό και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό διαφορετικά. Αλλά ακόμη και στην Ευρώπη πιστεύω απομένουν πολλά να γίνουν. Είδαμε τι έγινε με τα drones πάνω από το Παρίσι και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα τα απαραίτητα μέσα. Οπότε εσωτερικά θα πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας για το ζήτημα της αξιοπιστίας, του αξιόπιστου ε, υλικού και του αξιόπλου. Αυτό που λαμβάνουμε από τα κράτη μέλη ως προφορία αυτή τη στιγμή σε μια βάση δεδομένων ε, αποτελεί ένα καλό βήμα, πολύ ενθαρρυντικό. Φυσικά δεν θα μας αποκαλύψει τα κράτη μέλη όλες τους τις πηγές και ίσως αυτό να μην είναι καν και απαραίτητο. Αλλά μας βοηθά σε μια πιο πλήρη αξιολόγηση της γενικότερης εικόνας προσφερθεί και στην κοινή χρήση αυτή τη εικόνα ώστε να αποφύγουμε ε, υποθέσει όπω αυτή που συνέβη με τι μελισσιανέ αερογραμμέ στην 17. Ευχαριστούμε κύριο Γκαϊεύσκη. Καταρχά, να τονίσω ότι όλοι μας είμαστε επιβάτες ε, πτήσεων ανεξάρτητα από το που προερχόμεθα. Άρα τα θέματα ασφάλειας μας ενδιαφέρουν. Θέλουμε να ξέρουμε πώς έχει συμβεί ένα συγκεκριμένο ατύχημα. Και μάλιστα ένα, ένα αεροσκάφος εξαφανιστεί εντελώς από τα ραντάρ, όπως ε, το μαλαισιανό αεροσκάφος. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα μόνο για τη Μαλαισία, αλλά για όλους μας. Το επόμενο βήμα είναι όταν γίνει ένα ατύχημα να κάνουμε μια σωστή έρευνα για να δούμε γιατί συνέβη, πώς συνέβη. Και έχουμε στοιχεία επιβεβαιωμένα που αποδεικνύουν ότι ορισμένοι φορείς διερεύνησης ατυχημάτων δεν έχουν τις αναγκαίες γνώσεις για να κάνουν τέτοιες έρευνες. Αυτό ήθελα να σας παρουσιάσω. την ερώτηση για το ποιο τμήμα των κανονισμών του ΙΚΑΟ παραβίασαν οι Ρώσοι. Η κάθε χώρα μπορεί να κάνει έρευνες ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών της. Άρα δεν είναι η σωστή ερώτηση. Εάν ε, παρέβησαν κάποιο κανόνα, δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μία μόνομη διαδικασία. Κάθε χώρα κάνει μία έρευνα μέχρι το επίπεδο ικανότητάς της. Αν δεν μπορεί να κάνει σωστά την έρευνα, ζητάει συνεργασία άλλων χωρών. Γι' αυτό πολύ συχνά ο Καναδάς και οι Ηνωμένε Πολιτείε καλούνται να βοηθήσουν για να καταλήξουν κάποιες έρευνες. Δεν μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις για το Eurocontrol. Δεν είμαι ειδήμων για αυτά τα θέματα. Νομίζω ο κύριος Μπρένερ είναι ο αρμόδιος. Αυτά ευχαριστώ πολύ. are invited to conclude. Ο κύριος Μπρόκ για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για πολλούς λόγους. Πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με το θέμα αυτό και στα πλαίσια της Επιτροπής Μεταφορών, συνεργαζόμενοι. Γιατί είναι θέμα και μεταφορών, ιδίως από νομοθετικής άποψης. Υπάρχουν πολλοί εθνικοί εγωισμοί από ό,τι φαίνεται. Και λόγω και διαφόρων διαδηλώσεων και δράσης των συνδικάτων, και για όλους αυτούς τους λόγους η Κομισιόν απέσυρε τις φιλόδοξες προτάσεις της. Άρα δεν θα προχωρήσουμε. Αντίθετα θα επιβραδύνουμε από ό,τι αρχικά είχε προταθεί. Και από αυτά που λέει ο κ. Μπρένερ διαπιστώνω ότι οι τεχνικές δυνατότητες είναι πολύ πιο προθυμένες από ό,τι θέλουμε εμείς ως νομοθέτες να επιβάλλουμε. Αλλά επειδή είναι θέμα ασφάλειας δεν πρέπει να τίθεται το θέμα εάν ο καθένας πρέπει να διατηρήσει κάποιες ε, παραδοσιακές και τόσο αγαπημένε του αρμοδιότητες και δεν θέλει να εισαγάγει κάτι άλλο γιατί κάποιες θέσεις εργασίας, κάποιες αρμοδιότητες μπορεί να κινδυνεύσουν πρέπει να ισχύσει το πιο σημαντικό σήμερα το πρωί έμαθα ότι έπεσε ένα Airbus στην Νότια Γαλλία δεν ξέρω ακόμη τους λόγους δεν ξέρω, μπορεί να είναι θέμα τεχνικό, να μην έχει καμία σχέση με την κυκλοφορία. Μόλις το έμαθα, πριν από λίγα λεπτά. Βλέπετε λοιπόν ότι πάντα υπάρχει κίνδυνος και γι' αυτό πρέπει να κάνουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τη δουλειά, της, τη δουλειά τους επί των προτάσεων της Κομισιόν. Πρέπει λοιπόν να παρέμβουμε κι εμείς ταχύτατα να έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Μεταφορών και να τους ενθαρρύνουμε να έχουν φιλόδοξες προθέσεις. Διότι όλα αυτά τα επεισόδια σε περιοχές συγκρούσεων και όχι, αυτά που σχετίζονται με στρατιωτικά θέματα ή όχι, όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν και γι' αυτό στην επόμενη συνεδρίαση του Προεδρίου της ΑΦΕΤ, ε, δεν ξέρω πότε είναι αυτή η εβδομάδα ή την επόμενη, θα προτείνω να έρθουμε σε επαφή με την ε, Επιτροπή Μεταφορών για να δούμε πώς μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα και εντονότερα και ελπίζω να μπορείτε να μας βοηθήσετε και εσείς κύριε Μπρένερ και άλλοι εμπειρογνώμονες γιατί πρέπει να έχουμε μία ενιαία πολιτική μεταφορών. Αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαθα επαρκώς με την ασφάλεια. Και οπότε ο σέντε και ο σάφετ μας ενδιαφέρει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Να σας ενημερώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκλήθηκαν στην συνάντησή μας σήμερα διότι αναμφίβολα η συζήτηση που μόλις είχαμε προφανώς άπτεται και θεμάτων αρμοδιότητας της Επιτροπής Μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να συζητάμε από κοινού τα θέματα αυτά. Σήμερα ξεκίνησε η συζήτηση, πρέπει να συνεχιστεί μαζί με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Μεταφορών. Ο κύριος Μπρένερ μας έδειξε ένα συγκεκριμένο χάρτη όπου είδαμε πόσο περίπλοκη είναι η διαδρομή των πτήσεων των πολιτικών πτήσεων βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ περίπλοκα αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και περιοχές συγκρούσεων. Οι οποίες είναι κοντά μας εδώ, στα ανατολικά, στα νότια. Άρα χρειάζεται συντονισμός. Ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι η ασφάλεια είναι το πρώτιστο μέλημα. Οπότε κλείσαμε αυτό το θέμα της ε, συνεδρίασης. Θα συνεχίσουμε στις 3 με τα επόμενα θέματα της μέρης διάταξης.